Γεια σας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε στην ε, συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου Προεπολογισμού. Βλέπετε τις γλώσσες στο Cont News της συνεδρίασης, η οποία ε, μεταδίδεται απευθείας το διαδίκτυο. Θα περάσουμε αμέσω στο πρώτο σημείο που είναι η ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο την κυρία Μαριάν Τάισεν. Καλώς ε, καλωσορίσατε κυρία Επίτροπε. Με χαρά σας υποδεχόμαστε ε, παρουσία ε, του αρμοδίου μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου Ηλιάνα Ιβάνοβα που είναι αρμόδια για το συγκεκριμένο θέμα. Καλωσορίζω λοιπόν όλους τους προσκεκλημένους και όλα τα μέλη. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Ιβάνοβα. Madam Chair, Madam Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Συγητά, αξιότιμοι κύριοι Σε Μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι και πάλι εδώ για δεύτερη κατά σειρά εβδομάδα για να σα ε, παρουσιάσω το κεφάλαιο 3 6 ε, συγγνώμη, τη ετήσια έκθεση που καλύπτει την ε, κατηγορία του PDP 1β, Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή. Πριν να προχωρήσω στην παρουσίασή μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την ανοιχτή και επικοδομητική σχέση εργασία ε, που είχαμε μεταξύ μας και πάλι έχουμε συνεργαστεί αγαστά ολόκληρη τη χρονιά και όπως θα γνωρίζετε ο κοινωνικός τομέας ε, στις στα περισσότερα αν όχι όλα τα κατημέλη αντιμετωπίζει ε, αυξανόμενες πιέσεις άσχετα από την εθνικότητα, φύλο, παιδεία κτλ. Όλα τα μέλη της κοινωνίας μας θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται και να ζουν ειρηνικά. Όμως αυτό, η επίτευξη αυτού του απλού στόχου δεν είναι καθόλου απλή. Τα κονδύλια είναι λιγοστά πάντοτε και γι' αυτό και οι προεκκλήσεις για τα εθνικά συστήματα ώστε να είναι πιο, ε, ώστε μάλλον και το τελευταίο ευρώ που δαπανάτε να έχει όσο γίνεται μεγαλύτερο εφέ, ε, είναι πολύ μεγάλες. Θα ξεκινήσω δίνοντάς σας κάποια, κάποια στοιχεία από τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, εφόσον ε, έγινε, μπήκα σε λεπτομέρειες την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θα το κάνω και πάλι. Θα αναφέρω κάποιες στοιχείες για την νομιμότητα και την κανονικότητα. 8,1 ευρώ δαπανίσαμε 80% του συνόλου του τίτλου ε, για το PDP. Πρόκειται για πολιετή προγράμματα και τη διαχείρισή του είναι κοινή ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Κομισιόν. Όπως ανέφερα την περασμένη εβδομάδα, εκτιμόμενο περιθώριο σφάλματος, ο σύνολο ήταν 4,8%. Τα κύρια είδη σφάλματος είναι η μη, τα μη επιλέξιμα κόστη που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις ε, των ε, δικαιούχων 42%, ε, κρατικές προμήθειες 30% και μη επιλέξιμα project δραστηριότητες 28%. Έχουμε και ένα χωριστό τμήμα στο τέλος του κεφαλαίου που εκτιμά την απόδοση των project. Βρίσκουμε ότι ο σχεδιασμός του συστήματος απόδοσης, διαχείρισης απόδοσης ήταν πιο στεναρός για το περίοδο 2014 ας πούμε ότι οι έλεγχοι στα κράτη-μέλη, ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να ελέγξουν ε, τα στοιχεία περί αξιοπιστίας απόδοσης και η Κομισιόν ε, προβαίνει σε ελέγχους όταν υπάρχει ιδιαίτερα σημαντική υπολειτουργία ή ελλειπής επίτευξη των στόχων. Έχουμε λοιπόν τα project από την περίοδο μέχρι το 2013 τα οποία έπρεπε να ολοκληρωθούν αλλά μπορούμε να πούμε πως όλα τα project είχαν τους στόχους τους είτε πλήρως είτε μερικώς. Επίσης θα ήθελα να τονίσω κάποιες πτυχές για ε, ορισμένες ειδικέ εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν πέρσι στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων όπου εξετάζουμε περισσότερο την ετήσια έκθεση του 2016. Ήμουν επίσης μέλος για την έκθεση περί παιδείας στη, σημεριν... τη σήμερον εποχή η αξιοπρεπή παιδεία είναι πιο σημαντική από ποτέ και μια από τις θεμελιώδει αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πρόθεση της γνώσης προσφέροντας στους Ευρωπαίους πολίτες ευρεία πρόσβαση στην εκπαίδευση. Είναι ένας από τους πέντε τομείς όπου η στρατηγική 2020... Ε, της Ευρώπης 2020 έχει θεσπίσει συγκεκριμένους στόχους και η πρόοδο που έχει σημειωθεί είναι στοιχείο κλειδί τη δουλειά μα. Συμπέρασμά μα είναι ότι ενώ οι στόχοι για την παιδεία έχουν ληφθεί υπόψη στα επιχειρησιακά προγράμματα και project, έχουμε εντοπίσει κάποια μειονεκτήματα που μπορεί να επηρεάσουν την παρακολούθηση της απόδοσης. Και ενώ υπήρχαν κάποια προβλήματα, τα την περίοδο 2007-2013 για την περίοδο 2014 με 2020 παρατηρήθηκε σαφής βελτίωση. Το επόμενο θέμα που θα ήθελα σύντομα να σχολιάσω είναι ένα από το οποίο είναι ιδιαίτερα προσφυλές, προσφυλές, νεότητα και απασχόληση. Ξεκολουθεί να είναι σημαντική πτυχή αυτής ε, της ε, ε, αυτού του τομέα χρηματοδότηση της Ένωσης και ε, το μέλλον ε, των νέων στο χώρο εργασία είναι πολύ σημαντικό για την ευημερία ολόκληρη τη Ένωση. Νωρίτερα φέτος δημοσιεύσαμε τρίτη έκθεση για το ίδιο θέμα. Είχαμε την εγγύηση για την νεότητα και τη στήριξη τη Κομισιόν ε, για τι ομάδε δράση για του νέου. και τώρα μιλάμε για την εγγύηση για την νεότητα καθώ και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Επισκεφθήκαμε 7 κράτη-μέλη, όλα είχαν σημειώσει πρόβλημα πρόοδο στην εφαρμογή της εγγύηση για τους νέους και κάποια αποτελέσματα ήδη υπήρχαν, ωστόσο κανένα από τα κάτι μέλη δεν είχε εξασφαλίσει πως όλοι οι νέοι ε, στην απασχόληση ή στην ε, εκπαίδευση της, στην κατάρτιση δεν είχαν λάβει ε, κάποια προσφορά για εργασία εδώ και μήνες. Παρατηρήσαμε τις καλές πρακτικές στα κρατημέλη αλλά κυρίε και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, η δημοσίευση εκθέσεων επιδόσεων δεν είναι το τέλο, Ανέκαθεν έχω καταστήσει σαφέ ότι προσδίδουμε μεγάλη σημασία σε άλλε μορφέ επικοινωνία, εφόσον θέλουμε να περάσουμε τα μηνύματά μα στου διάφορου φορεί. Και την αρχή αυτή τη θέσαμε σε εφαρμογή νωρίτερα φέτο, καθώ ε, έγινε μια, διοργανώθηκε μια διάσκεψη για την απασχόληση των νέων φέτο μετά από τη δημοσίευση τη έκθεση πρόοδου και με χαρά ε, διοργανώσαμε αυτήν την διάσκεψη εδώ στο Κοινοβούλιο μαζί με την εξαίρετη συνεργασία της Κομισιόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου που παρακολούθησαν και συνέβαλαν σε αυτή την εκδήλωση. Να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο Τάισεν και την ομάδα της, το επιτελείο της, για την προσήλωσή της στο θέμα. Και ε, εδώ συμμετείχαν πάνω από 300 συμμετέχοντες που παρακολούθησαν και παρακολούθησαν επίσης πολύ ε, στο ίντερνετ την απευθεία αναμετάδοση. Κύριε, κύριε εισηγητή, κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι πάντοτε μεγάλη μου χαρά να έρχομαι στην Επιτροπή και ελπίζω πως τα σχόλιά μου θα είναι μια υποφελή ε, συμβολή στη συζήτησή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ιβάνοβα και ευχαριστώ για την αφοσίωσή σας στο θέμα της απασχόλησης και ιδιαίτερα στο θέμα της απασχόλησης των νέων. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο και ε, σας ακούμε μεγάλη προσοχή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, αξιότιμη κύριε Σιγητά, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρία Ιβάνοβα, κυρίες και κύριοι. Στην αρχή της θητείας μας δεσμευθήκαμε για την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτή θα συμβάδιζε με τη βελτίωση των ζώων των πολιτών. Η Ευρώπη θέλουμε να έχει ένα κοινωνικό τριπλό α, α ανάπτυξη δίκαιη, ισορροπημένη, με δημιουργία θέσεων ε, εργασίας ε, ποιοτικών, καλύτερη κοινωνική προστασία και κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Έχουμε λάβει μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα για να το επιτύχουμε αυτό ήδη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων τον ε, παρουσιάσαμε την Άνοιξη που πρόσφατα διακήρυξαν και τα τρία ε, θεσμικά όργανα στο Γκέτεμπεργκ, στον ε, Σύνοδο Κορυφής για τον Κοινωνικό Πυλώνα. Θέλουμε ένα πλαίσιο για μια αγωνιστική, δυναμική αλλά και δίκαιη οικονομία έτσι ώστε να πετύχει και να διαφυλαχθεί το κοινωνικό μας μοντέλο. Χωρίς κοινωνικό ντάμπινγκ το έχει πει αυτά και ο πρόεδρο Γιούνκερ ε, το Σεπτέμβριο στην ομιλία του για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, εργαζόμαστε ε, προ τη μείωση τη ενέργεια των νέων. Το καλοκαίρι, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, επέκτηναν κατά 1,2 δισεκατομμύρια το αντίστοιχο πρόγραμμα για την περίοδο 17 ε, 20 δείχνοντας ότι υποστηρίζουμε τις πολιτικές προτεραιότητες ε, για να καταπολεμήσουμε τις συνέπειες οικονομικής κρίσης και οι άνθρωποι που επλήγησαν να επανέλθουν στην εργασία τους. Επίσης, για την απόσπαση των εργαζομένων να επιδιώκουμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία της αγοράς, την προστασία των εργαζομένων και τους ίδιους κανόνες ε, παιχνιδιού για τους επιχειρηματίες. Χαιρόμαστε ε, για τις επιτυχίες ε, σχετικά που σημείωσε η Εστονική Προεδρία και ε, την εντολή των δύο διαπραγματευτών, μάλλον των δύο εισηγητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αρχίσουν διαπραγματεύσεις και ελπίζω γρήγορα να προχωρήσουμε στους επόμενους μήνες. Μια πολιτική όμως για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει σωστά να εφαρμόζεται και συγκεκριμένα επιτόπου και εδώ θα έρθουμε να γεφυρώσουμε την πολιτική μας στη θεωρία με την πραγματικότητα. Είναι πολύ θετικά τα σημεία. Αυξάνεται η ανάπτυξη παντού στην Ευρώπη πάνω από 2% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2,2% στις ε, χώρες της Ευρωζώνης. Η ανεργία είναι χαμηλότερη στις τελευταίες εννέα ετίας, σχεδόν 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν όπου απασχολούνται προφανώ 8 εκατομμύρια εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια τη παρούς θητείας. Επίσης, συνεργαζόμαστε με του ε, τέρους μα τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε τα χρήματα ε, και οι πόροι μα να δαπανώνται με τρόπο αποτελεσματικό και σωστό. Και χαίρομαι που το ελεγκτικό συνέδριο και φέτο, αντανακλά ε, στις εκθέσει του τη σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει για να πλουστεύσουμε και να εξυγχρονίσουμε του οικονομικού κανόνε, έτσι ώστε και ο έλεγχο να γίνεται με σωστό τρόπο στα πλαίσια της οικονομικής, κοινωνικής και δαφικής συνοχής για πέμπτη συνεχή χρονιά διαπίστωσε στο συνέδριο μείωση του σφάλματος στη συνοχή. Το 2016 είναι στο 4,8% ενώ το 2015 ήταν 5,2% επιπλέον για τις πληρωμές για, για πρώτη φορά εξέδωσε δικαιολογημένη ε, γνωμοδότηση το ελεκτικό συνέδριο και αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε προχωρήσει σε ό,τι αφορά την νομιμότητα και τη, το τυπικό των διαδικασιών. Το 2016 λοιπόν είναι το τελευταίο έτος όπου ε, η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο έχει ελέγξει την προηγούμενη προγραμματική περίοδο για τελευταία φορά, 2007-2014. Ελπίζουμε και για την επόμενη προγραμματική περίοδο να συνεχιστεί η ε, θετική τάση στις επόμενες χρήσεις. Το Ελεκτικό Συνέδριο συμπίπτει στις εκτιμήσεις του με τις υπηρεσίες μου για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. 3,9% των σφάλμα για το κοινωνικό ταμείο για τις πληρωμές του 2016 όλα τα ε, οικονομικά εργαλεία που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης ε, συνολικό σφάλμα ήταν στο 3% λαμβάνοντας υπόψη ε, οικονομικές διορθώσεις οι υπηρεσίες μου υπολογίζουν το υπολοιπόμενο σφάλμα για το 2016 να είναι μόλις 0,8%. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε όταν μιλούμε για σφάλμα ότι δεν πρόκειται για απάτη η διαφθορά, η αναποτελεσματικότητα, η διασπάθηση, αλλά μάλλον για τα χρήματα που καταβλήθηκαν και δεν απορροφήθηκαν ε, ή δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους. Αυτά όλα δεν είναι τυχαία. Ε, είναι καρπός των προσπάθειών μας η απλούστευση και εξυγχρονισμό του συστήματος. Για πέμπτη συνεχή χρονιά λοιπόν επιβεβαιωνόμαστε στην προσέγγιση μας. Το Ελεκτικό συνέδριο δεν έχει ε, εντοπίσει μετρήσιμο σφάλμα για ε, την προηγούμενη τετραετία ούτε για φέτος. Μια πρόσφατη μελέτη απλούσευσης δείχνει ότι 35% των πόρων του κοινωνικού ταμείου απορροφούν ε, σύμφωνα με τις επιλογές ε, απλουστευμένου κόστους σε σύγκριση με ένα 7% που ίσχυε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Επιπλέον, ε, τα επιχειρησιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κατά την πλειονότητά τους χρησιμοποιούν επιλογές απλουστευμένου κόστους, ενώ Αυτό ισχύει για, τα μισά κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου. Για την περίοδο 2014-2020 και τα αντίστοιχα ΕΣΠΑ είναι γεγονός ότι υπήρξε μια δυστοκία στην αρχή. Άργησε να εγκριθεί ε, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μόλις το Δεκέμβριο του 2013 το τον οι νομοθέτες, γι' αυτό άρχισε να ξεκινήσει κιόλας. Επίσης και ο κανόνας νήσιν 3 οδήγησε σε αύξηση απειθαρχίας σε κάποιες εθνικές διοικήσεις όταν εκλήθησαν να τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Και επίσης μερικά από τα νέα στοιχεία που έχουμε εισαγάγει ε, στη νέα περίοδο, την προγραμματική 2014-2020, ε, όπως η απέτηση να οριστούν ελεκτικές αρχές και ορισμένες ε, διατάξεις της εκ των προτέρων ε, οδήγησαν σε καθυστερήσεις ε, της εθνικές δίκης. Ε, ωστόσο, σήμερα διαπιστώνουμε ότι το 96% ε, των αρχών που διαχειρίζονται τους πόρους του Κοινωνικού Ταμείου έχουν οριστεί. Και στις εκθέσεις πρόοδου και στις εκθέσεις εφαρμογής φαίνεται ότι σχεδόν το σύνολο των των προτέρων όρων τηρούνται αυτή η εξάντε αιρεσιμότητα επιπλέον υπάρχει ισχυρότερο επενδυτικό περιβάλλον και κίνητρα για επενδύσεις υψηλής ποιότητας. Επίσης έχουμε και σαφή σημεία ότι θα επιταχυνθεί η εφαρμογή, η υλοποίηση το επόμενο διάστημα. Από το 20% που ήταν το τέλη του 2016 έχει αυξηθεί ήδη στο 40% φέτος ο ρυθμός έγκρισης των προγραμμάτων και των έργων που εμπίπτουν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Κύριε Σεγητά, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως γνωρίζετε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το βασικό εργαλείο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίζει τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Τώρα που έχουμε ξεπεράσει τη μισή θητεία μας, ε, φαίνεται ότι αποδίδει στην πράξη, ότι είναι κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης για ευάλωτες ομάδες που υπέστησαν τις τη της κρίσης. Επίσης ήταν αξιόπιστη πηγή επενδύσεων σε περιόδους ασταθών χρηματαγορών και αλλαγών στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Επίσης έχει αποδειχθεί αρκετά ευέλικτο έτσι ώστε να υποστηρίξει και να απαντήσει στην ε, κρίση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού. Πάντα μαζί με τα ταμεία προς τους πιο ευάλωτους απόρους που έχουν υποστηρίξει ε, ετούντες άσυλο, μετανάστες και άλλες ευάλωτες ομάδες. Πάντα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχουμε αποτελέσματα στη στήριξη των ανέργων, ε, των ανθρώπων χωρίς δεξιότητες, ανειδίκευτων, εκείνων που χρειάζονται αλλαγή ε, στην εκπαίδευσή τους, μετακπαίδευση για να βρουν εργασία. Να σας δώσω μερικά στοιχεία. Στο προηγούμενο πρόγραμμα, προγραμματική περίοδο εννοώ, και μέχρι τα τέλη του 2014 τουλάχιστον 9,4 εκατομμύρια ε, άνθρωποι μπήκαν στην αγορά εργασίας. Πάνω από 300.000 ε, αυτοαπασχολούμενοι μεταξύ αυτών και 8,7 εκατομμύρια ε, έλαβαν πιστοποίηση ή έλαβαν κάποιο αποδεικτικό ότι ε, ε, έχουν κάποια κατάρτιση από το Ταμείο Κοινωνικό. Για την επόμενη περίοδο 2014-2020 έχουμε επίσης θετικά στοιχεία και τους πρώτους καρπούς. Η πρώτη στρατηγική έκθεση που θα δημοσιεύσουμε τις επόμενες εβδομάδες δείχνει ότι μέχρι το τέλος του 2016 η ε, πρωτοβουλία για τους νέους και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστήριξαν 7,8 εκατομμύρια πολίτες. Από το 2013 μέχρι σήμερα είναι 2 εκατομμύρια λιγότεροι οι άνεργοι στην Ευρώπη. Και μειώνεται ο αριθμός των νέων ανέργων στην Ευρώπη συνεχώς. Μάλιστα με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι θα ανέμενε κανείς δεδομένου του μακροοικονομικού πλαισίου. Αυτό δείχνει σαφώς την προστιθέμενη αξία της συγκεκριμένης πολιτικής. η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων που είναι το βασικό εργαλείο που έχουμε για να βρουν οι ε, νέοι ε, εργασία, εκπαίδευση, κατάρτιση και μάλιστα στις πιο ευάλωτες περιφέρειες έχει υποστηρίξει άμεσα πάνω από 1,6 εκατομμύρια νέους και από τον Ιανουάριο του 2014 πάνω από 18 εκατομμύρια νέοι έχουν μπει σε αυτά τα προγράμματα. Ενώ 11 εκατομμύρια ε, δέχτηκαν μια προσφορά για εργασία, μαθητεία, άσκηση ή συνέχισαν ε, την εκπαίδευσή τους. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, οι προσπάθειές μας εξακολουθούν να αποφέρουν ε, Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά το νομότυπο και το νόμιμο της διαχείρισης και επικεντρωνούμε τα κονδύλια μας σε βασικές πολιτικές και στόχους που έχουμε συμφωνήσει από κοινού. Ωστόσο, το έργο μας δεν σταματά εδώ και στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετές του δημοσιονομικού πλαισίου έχουμε υποβάλει φιλόδοξες προτάσεις για περαιτέρω απλούστευση των κανόνων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Θέλουμε να αυξήσουμε ας πούμε σε 100.000 ευρώ το ε, κατόφλι για κάποια υποχρεωτικά σχήματα που υπακούν σε κάποιους όρους και προϋποθέσεις. Είμαι επεπισμένη ότι τέτοιου είδους μέτρα ε, μαζί με την ενίσχυση του προγράμματος για την επόμενη περίοδο θα μας βοηθήσει για να βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω την αποτελεσματική ε, εφαρμογή του Κοινωνικού Ταμείου της Εγγύησης Νεολαίας και να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο στους λογαριασμούς. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την επόμενη προγραμματική περίοδο θα πρέπει να προβληματιστούμε, να απλοποιήσουμε ριζικά ε, τους κανόνες και ε, τα προβλήματα που έχουμε ε, δει παντού. Η απλοποίηση μας επιτρέπει να ε, δαπανούμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα χρήματα των φορολογουμένων. Και άρα να πιάνουν τόπο τα κονδύλια αυτά και να εμφανίζουν μια προστιθέμενη αξία ε, της Ευρωπαϊκή Ένωση στα μάτια των πολιτών, βελτιώνοντας τη ζωή τους. Αυτό θα πρέπει να κυριαρχήσει στη συζήτησή μας για το επόμενο ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο ε, υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή οικονομία, κοινωνική οικονομία της αγοράς ε, με τον κοινωνικό πυλώνα τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που ε, ανακηρύχθηκε πρόσφατα στο Σύνοδο Κορυφής για τα κοινωνικά θέματα στο Γκέτεμπορ. Η κανόνα μας θα πρέπει να είναι καλή, ευέλικτη, να εξυπηρετούν το στόχο και να συναντούν την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στην συμμόρφωση και την απόδοση και τις επιδόσεις. Θα πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι και τα κράτη-μέλη να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, έτσι ώστε οι θεμελιώδεις αρχές του κοινωνικού πυλώνα να γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα για όλους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ και πάλι για σας και το επιτελείο σας για τις απαντήσεις. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δουλειά που κάνετε και πάρα πολύ ε, χρήσιμο για μας να έχουμε τις γραπτές απαντήσεις για να τις χρησιμοποιούμε στην ανταλλαγή απόψε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσέλερ, τον εισηγητή μας. Παρακαλώ. Ähm, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη κυρία Ιβάνοβα και κυρία Τάισεν που σας γυρίζω την πλάτη. Έχει να κάνει τώρα με τη διάταξη της αίθουσα και το πώς καθόμαστε. Δεν έχει καμία σχέση με αγένεια, το αντίθετο μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ιβάνοβα και τους συνεργάτες της ε, για την ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για το 2016 που αποτελεί τη βάση έτσι ώστε να χορηγήσουμε την έκθεση από την απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Οικονομικό έτος 2016 και να εκπονήσουμε την αντίστοιχη έκθεση. Κυρία Τάισεν, αξιότιμη κυρία Επίτροπε, θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς και το γενικό σας διευθυντή και τους συνεργάτες σας που απαντήσατε στις 48 μας ερωτήσεις, ερωτήσεις που σας είχαμε διαβιβάσει με πάρα πολύ υλικό, με αριθμούς και στοιχεία τεκμηριώνονται πράγμα που βοηθάει και βελτιώνει και την έκθεσή μας. Πρέπει να τονιστεί αυτό που είπαν και οι δύο κυρίες και η κυρία Ιβάνοβα και η κυρία Τάισεν, ότι και πάλι καταφέραμε το ποσοστό σφάλματος να μειωθεί κατά την εφαρμογή ε, και την εκτέλεση των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και άλλων διαφορετικών ταμείων έχει φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο το οποίο είναι κοντά ε, στο 2% που είναι το όριο του στατιστικού σφάλματος. Άρα ε, Τώρα πλέον δεν συζητάμε τα τυπικά για τη συμμόρφωση και τα λοιπά, αλλά τα ουσιαστικά για το τι κάνουμε ακριβώς με τα διορθωτικά ταμεία και τι θέλουμε να επιτύχουμε. Μπορούμε να το αποδείξουμε πλέον. Και επίσης πίσω από τους αριθμούς, που κρύβονται πίσω από τους αριθμούς ε, ανθρώπινες ζωές και μοίρες και πεπρωμένα, ε, αποδεικνύουμε ότι ε, γίνονται προσπάθειες στον κοινωνικό τομέα που εξαρτώνται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το είπε και η κυρία Επίτροπος, σε ό,τι αφορά την απασχόληση αυτή τη στιγμή, διαπιστώνουμε θετική εξέλιξη. Το 2007 η τελευταία έκθεση συνοχής ε, λέω ότι η απασχόληση έχει φτάσει στο 71% ενώ η ανεργία από 11% στο 8,6% έχει πέσει. Δεν χωράει καμία αφιβολία ότι αυτό είναι επιτυχία που έχει να κάνει και με κάποια μακροοικονομικά φαινόμενα. Ωστόσο, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών υπάρχουν πολύ διαφορετικοί διαφορετικές ε, πραγματικότητες και αποτελέσματα. Υπάρχουν χώρε με πολύ χαμηλή ενεργεία και υψηλή η απασχόληση και χώρες ε, που γνωρίζουν ακριβώ το αντίθετο. Πολύ δε περισσότερο που εκεί είπατε εσείς κύριε Επίτροπε και εσείς και οι συνεργάτε σα στις γραπτές απαντήσεις αν υπάρχουν νέε προκλήσεις για την κοινωνική πολιτική τα τελευταία χρόνια ακριβώ έχουν έρθει στην Ευρώπη πολλοί ως πρόσφυγες, μετανάστες ή αιτούντες άσυλο οι οποίοι πολύ συχνά δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο των προσόντων και δεξιοτήτων που απαιτεί η αγορά μας. Πολλές φορές είναι μέχρι και αναλφάβητοι ή τουλάχιστον δεν γνωρίζουν τις γλώσσες ε, που μιλούνται στις χώρες μας. Και εκεί έχουμε ζητήματα και κοινωνικής πολιτικής που χρειαζόμαστε ένα νέο προσανατολισμό των διευθυντικών ταμείων για να βοηθήσουν την κατάσταση. Διάφορε πηγέ και το ελεκτικό συνέδριο μεταξύ αυτών λέγουν ότι τα προσόντα και οι δεξιότητες που προσφέρονται και παρέχονται δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που ζητάει η αγορά. Και αυτή ε, η ε, αναντιστοιχία αποτρέπει την περαιτέρω πρόεδρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δέχεται αυτό, αλλά λέει ότι έχει αλλάξει και η αγορά ο, ο τρόπος ε, πρόσληψης, η ευελιξία, η έλλειψη δυνατοτήτων ανέλυξης ε, δεν είναι μόνο η αντιστοιχεία των προσόντων. Τι ε, συστάσεις θα μπορούσε να απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρωζώνη στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και πώς αξιολογεί τις μεταρρυθμίσεις που κάνουν τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο. Θυμάμαι ακόμα στη δεκαετία του 90 στη Γερμανία μετά την επανένωση την ανεργία που ήταν αρκετά ψηλότερη από ό,τι είναι σήμερα. Ελήφθησα μέτρα ενίσχυσης της αγοράς εργασίας και μόνο στο Βερολίνο ε, ε, έκαναν ε, εκπαίδευση για ξέρω εγώ 200 τοπογράφους αλλά δεν χρειαζόταν τοπογράφους στο Βερολίνο ε, οι στατιστικές έτσι τους βγάλαν από την ανεργία αλλά τους έστειλαν σε μια εκπαίδευση και μια κατάρτιση που δεν είχε επαγγελματικέ προοπτικές. Ή... Ε, Κανένα ορίζοντα να βρουν κάποτε δουλειά. Αυτά λοιπόν υπάρχουν ε, θέματα που πρέπει να συζητήσουμε και στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Η Αρχή Ελέγχου του Προπολογισμού επανειλημμένα έχει ζητήσει από τη Γενική Διεύθυνση να κάνει προτάσεις για τις συστάσεις αναχώρα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στις αιτήσεις εκθέσεις ε, πεπραγμένων. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εμεί από το Κοινοβούλιο θα επιθυμούσαμε από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης να κάνετε προτάσεις για τις συστάσεις αναχώρα. Δεν είναι τίποτα απόρριτο αυτό. Θα πρέπει να είναι τμήμα της δημόσιας συζήτησης. Στα μέτρα κοινωνικής πολιτικής κυριαρχεί η πρωτοβουλία για την νεολαία. Πάνω από 700.000 νέοι έχουν υποφεληθεί, εκ των οποίων η μισή περίπου προχωρούν σε μετεκπαίδευση, κατάρτιση, άσκηση, μαθητεία, πρόσληψη, συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα. Αυτό που έχει για μένα σημασία είναι να διατηρηθεί αυτό το μέσο και να, να είναι βιώσιμο για να μην ξεφουσκώσει αυτή η προσπάθεια. Όπως σας είπα το προηγούμενο Παράδειγμα, να μην εκπαιδεύουμε τον κόσμο για δουλειές που δεν υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να γεννάμε φρούδες ελπίδες ε, στα μάτια των νέων με κάποια εκπαίδευση και, και κατάρτιση που δεν θα καταλήγει πουθενά παρά μόνο στο πεζοδρόμιο ξανά. δεν μου αρέσει και ο τρόπος που απορροφώνται τα κονδύλια, όπως και στα κονδύλια για τα περιφερειακά ταμεία και σε άλλα διαρθωτικά ταμεία. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ερχόμαστε να διαπιστώσουμε ότι μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου έχουν απορροφηθεί μόλις 30% των κονδυλίων. Και το 40% είναι προκαταβολές και συνολικά το δούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πανευρωπαϊκά δεν είναι καλύτερη κατάσταση. Μέσα Οκτωβρίου ήταν να απορροφηθεί μόνο 5,1% των διατεθειμένων κονδυλίων και τα περισσότερα πάλι ήταν προκαταβολές. Μία εξήγηση για τη χαμηλή απορρόφηση, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι ο χρόνος παλαιότερα ήταν νησιν 2, έχει γίνει τώρα νησιν 3 για την απορρόφηση. Επίσης, στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο Είχαμε μεγάλες ε, καθυστερήσεις και καθυστέρηση στην έναρξη. Και εξ όσων γνωρίζω, τώρα πολλές διαχειριστικές αρχές διαχειρίζονται ακόμα προγράμματα της τελευταίας περίοδου, παρόλο που τον ΙΣΥΝ 3 έχει εκπνεύσει, θεωρητικά. Αν συνεχίσει έτσι αυτή η εξέλιξη, υπάρχει ένας κίνδυνος και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο που έτσι κι αλλιώς ξεκίνησε πάρα πολύ αργά να έχουμε μετακύληση και παράταση του προγράμματος της εκτέλεσης στην επόμενη. Και το θέμα της επιτάχυνσης πραγματικά τίθεται με πολύ οξύ τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι φρονεί σχετικά. Μήπως θα έπρεπε να επανέλθει αυτό το νησιν 3 να γίνει νησιν 2 για να μην πω νησιν 1. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει επιτάχυση στην απορρόφηση και την εκτέλεση των ε, πόρων από το κοινωνικό ταμείο. Προσωπικά θα έλεγα ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα έχω τις επιφυλάξεις μου. Αλλά κάπως θα πρέπει να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να δραστηριοποιηθούν λίγο περισσότερο για την εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων τους. Στην ερώτηση παρθμών 25 διαβιβάζουμε στην Κομισιόν κάποιες συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου για τους νέους και τους ανθρώπους που είναι εκτός αγοράς, για το κόστος και τα χρήματα που είναι στη διάθεση των κρατών μελών. Δεν έχουμε πάντα στοιχεία. Ακούμε τι δίνει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπάρχει συνυπευθυνότητα, συγχρηματοδότηση. Τι γίνεται με τα κονδύλια που βάζουν τα κράτη-μέλη. Πώς μπαίνουν οι νέοι στην αγορά εργασίας. Επίσης ε, δεν έχουμε τα στατιστικά στοιχεία που χρειαζόμαστε. Όλες αυτές τις τάσει του ελεγκτικού συνεδρίου μπορεί να απευθύνονται στα κράτη-μέλη, αλλά ο δικός μας συνομιλητής είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς συνεργάζεται τώρα με τα κράτη-μέλη για να έχουμε βελτίωση της κατάστασης. Κάτι άλλο που είπατε εσείς κυρία Επίτροπη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση έχει κάπως ε, ενηλικιωθεί αυτό το ταμείο. Απαντάει η Κομισιόν στην ερώτηση του Κοινοβουλίου μήπως μπορούν να μειωθούν τα κονδύλια από εκεί. όχι. Γιατί ε, απορροφώνονται πολλά κονδύλια από το ταμείο αυτό ακόμα. Μήπως τότε να αλλάξει νομική βάση. Αυτό που έχω δει μέχρι τώρα τα τελευταία χρόνια από αιτήσει από πλευράς κρατών μελών για το Ταμείο Καταπολέμησης της Παγκοσμιοποίησης για μέτρα ε, στήριξης των έργων μετά από μαζικές απολύσεις. Πολλές φορές δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με την παγκοσμιοποίηση. Όταν ιδρύθηκε το Ταμείο είχε σκοπό να βοηθάει τις περιφέρειες όπου μεταγκαθίστανται επιχειρήσεις, φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πηγαίνουν κάπου αλλού ε, λόγω της παγκοσμιοποίησης και το ποσοστό των απολύσεων, ε, ο αριθμός ε, είναι μεγάλος, πάνω από 500 εργαζόμενοι. Τώρα στο εμπόριο όταν γίνεται λόγος για χρήματα που πηγαίνουν για μαζικές απολύσεις εργαζομένων στο εμπόριο, επαναλαμβάνω. Μα τι σχέση έχει αυτό, έχει ακόμα σχέση με την παγκοσμιοποίηση ή μήπως με τις ε, κατατόπους εξέλιξη της οικονομίας. Εγώ θα ήθελα να υποστηρίζουμε περιφέρειες που πλήττονται από την μαζική και ξαφνική ανεργία λόγω παγκοσμιοποίησης. Αν θέλετε να τα χρησιμοποιείτε και αλλού, ε, πρέπει να αλλάξει νομική βάση όταν έχουμε πολλές και μαζικές απολύσεις. Και να προσθεθεί και η διαδικασία εφόσον αλλάξει νομική βάση. Είχατε την καλοσύνη στο σημείο 11, στην ερώτηση 11 δηλαδή, να απαντήσετε σε αυτό το θέμα και να μας δώσετε τα στοιχεία που σας ζητούσαμε. Πάντα για τις μαζικές απολύσεις και κατά πόσο ενημερώνονται εκ των προτέρων οι εργαζόμενοι. Εδώ ε, απέχουν τα στοιχεία ε, από, ε, έχουμε μια ευρία γκάμα από 19% μέχρι 88% για τα ελακτικά συστήματα και τα συστήματα διοίκησης 23 προγράμματα λέτε έχετε επιφυλάξει για αυτά 5 στη Γερμανία η Ιταλία και η Ισπανία ήταν πάνω από δύο χρόνια σε μια επιφύλαξη. Γιατί δεν διεκπεραιώνονται αυτά πιο γρήγορα. 200 εκατομμύρια ευρώ ανέκτησε κονδύλια Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016 από την Ιταλία και την Ισπανία της περίοδου 2000-2006. Γιατί χρειάστηκε μια δεκαετία για να τα πάρετε πίσω αυτά τα λεφτά. Γιατί μας απαντάτε είναι πολύ περίπλοκη η διοίκηση σε κάποια κράτη-μέλη και η μηχανοργάνωση και το καλύτερο σύστημα μηχανοργάνωσης έχει τεχνικές δυσκολίες και νομικές. Ποιες είναι αυτές οι νομικές και τεχνικές δυσκολίες. Πρόσφατα ε, είχα συνομιλία στη Γερμανία με πολλές διαχειριστικές αρχές που ε, κάνουν αυτή τη δουλειά εδώ και πολλές προγραμματικές περιόδους και ε, είπε ότι έχει διωγγωθεί τόσο πολύ η διαδικασία έγκρισης ενός έργου που δυσκολεύονται και αυτές οι ίδιες οι αρχές που κάνουν αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια και τόσες προγραμματικές περιόδους. Ιδιαίτερα η εξάντα αιρεσιμότητα είναι κάτι το οποίο επικρίνουν σπόδρα και θα πρέπει να το ξαναδούμε με τις διαχειριστικές αρχές που στο κάτω-κάτω είναι ο ημάντας μεταβίβασης για μας έτσι ώστε τα ταμεία τα διαρθρωτικά και το κοινωνικό να ε, εκτελούνται σωστά και να βελτιώνεται το σύστημα και στην ανάθεση των έργων. Αλλιώς κινδυνεύουμε να έχουμε περαιτέρω καθυστέρηση στην απορρόφηση και δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι μέχρι το τέλος της προγραμματικής περίοδου μόλις το 35% του κόστους θα έχει υπολογιστεί με το νέο απλουστευμένο σύστημα η κυρία Τάισεν το χαρακτήρισε αυτό πρόοδο. Δεν μπορεί να επιταχυνθεί η πρόοδος. Ένα άλλο προσφυλές μας θέμα στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού είναι τα χρηματοδοτικά μέσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει πάντα ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και ο σκιώδης προϋπολογισμός πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Κοιτάξτε όμως λίγο παρακαλώ ε, τους γαλαξίες που έχουμε στην αρχιτεκτονική, το λέτε αυτό στη σελίδα 4, τον οικονομικό διαφάνεια, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από όλα αυτά τα ανεφελώματα. Και συμφωνώ με τον Επίτροπο Oettinger, αρμόδιο για τον προπολογισμό, ότι όλα αυτά ε, τα πληθωριστικά μέσα που έχουμε ε, που ξεχυλίζουν εκτός προϋπολογισμού θα πρέπει να επανέλθουν κάτω από την ενιαία στέγη του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και με χαρά, κυρία Επίτροπε, θα σας ακούσω να συμφωνήσετε αν συμφωνείτε μαζί μου, που δεν είμαι μόνο εγώ αυτός που τα λέει. Τι θα γίνει με τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, θα οδηγήσουν σε σαφή αξιόλογη βελτίωση ε, της απασχόλησης αν δεν τα διαχειρίζεται αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και με περηφάνεια δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μέχρι ε, τέλους του 2016 έχει δώσει 62.000 ε, μικροδάνεια λέγονται αυτά με μικρές ποσότητες μέχρι 1.100 ευρώ. Αν τα συνυπολογίσουμε όμως συνολικά είναι 6 εκατομμύρια ευρώ τα τραπεζικά έξοδα που πηγαίνουν ε, ως προμήθεια στην τράπεζα και τα χάνει η κοινωνική πολιτική. Αυτά εισαγωγικά. Σταματώ εδώ το σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Επίτροπε, όπως βλέπετε ο εισηγητής μας είναι πάρα πολύ σχολαστικός με πρόσθετες ερωτήσεις, οπότε θα σας δώσω το λόγο πριν περάσουμε στα μέλη ε, της ομάδας μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα απαντήσω στα Ολλανδικά, αφού έχω και διερμηνία. Και πραγματικά ε, θυμάμαι από παλιά την εξαιρετική ποιότητα των διερμηνέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την προηγούμενη ιδιότητά Ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι, πραγματικά είναι πολλά τα χρήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοδομητική σας ε, στάση και την καλή συνεργασία που είχαμε. Νομίζω ότι γενικά μπορώ να πω ότι το λέει και ο εισηγητής ότι έχει βελτιωθεί η ανεργία ε, μειώνεται, σιγά σιγά πραγματικά μειώνεται, αλλά πραγματικά υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών πολύ μεγάλες διαφορές. Είναι γεγονός αυτό σε ορισμένε χώρε έχουμε πλήρη απασχόληση, ενώ σε άλλε χώρες πάνω από 20% ανεργία. Και παρά όλη την πρόεδρο που έχουμε επιτύχει και την οικονομική μεγέθυνση ε, και τις μεταρρυθμίσεις, υπάρχουν άνθρωποι ε, που δεν εποφελούνται από την ε, ανάπτυξη που επιστρέφει και όπως είπε και ο εισηγητής έχουμε και νέα προβλήματα. Ε, Ήρθαν ε, μεγάλες προσφυγικές ροές, μεγαλύτερες από ό,τι ποτέ, αλλά έχουμε και την παγκοσμιοποίηση που έχει αφήσει πληγές και η ψηφιοποίηση που είναι πολύ μεγάλη πρόκληση και ανησυχία για μας και θα πρέπει πραγματικά να το μεταφράσουμε ε, στο επόμενο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Να υπάρχουν αρκετά χρήματα για την κοινωνική πολιτική, να είναι ορατά, να πιάνουν τόπο και να συνδέονται καλύτερα από ποτέ με τους ευρωπαϊκούς μας στόχους. Γιατί πραγματικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια να δημιουργούν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και εδώ σκέφτομαι τις μεταρρυθμίσεις που ζητούμε από τα κράτη-μέλη στις συστάσεις αναχώρα για το ευρωπαϊκό εξάμεινο να υπάρχει και συμμετοχή των ευρωπαϊκών κονδυλίων και ταμείων, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και άλλα ταμεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Μιλήσατε για τις προσφορές εργασίας ε, και τις ε, ε, πρωτοβουλίες για την νεολαία και την εγγύηση για την Ελλάδα λέτε ότι δεν είναι πάντα πολύ καλή ποιότητα οι προτάσει που του γίνονται. Αυτό πώ μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Και τα κράτη-μέλη. Πολλέ φορέ δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε ε, και να το αξιολογήσουμε. Το ξέρω ότι δεν είναι της καλύτερης δυνατή ποιότητα. Ε, θα αναπτύξουμε κάποιου δείκτε για να τα παρακολουθούμε. Αλλά για του needs, τους νέου που είναι εκτό εκπαίδευση, κατάρτιση μαθητεία, ε, ή εργασίας ε, είναι τελείως ξεκρέμαστοι. Δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Και ε, καλό είναι να έχουμε αυτές τις προσπάθειες, τουλάχιστον να καταγράφονται κάπου και κάποια στιγμή να βρίσκουν δουλειά. Δεν λέει τίποτα το ελεγκτικό συνέδριο για το πώς θα βρούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο μακριά από την εργασία, που είναι πραγματικά ε, απαγκιστρωμένοι από το σύστημα. Αυτοί είναι πιο δύσκολοι να βρεθούν, να καταγραφούν. Έχουμε εμεί μια κλασική δομή ε, που είναι ο ΑΕΔ, ξέρω εγώ, ή κάποιοι οργανισμοί απασχόλησης και ε, εργατικού δυναμικού κλπ. Αυτούς δεν τους βρίσκουν πουθενά, δεν είναι καταγραμμένοι σε στατιστικές θα πάμε να τους βρούμε εκεί που βρίσκονται και που κάθονται ε, άεργοι στη μέση του δρόμου γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν και να τους επαναφέρουμε σε ένα δρόμο που θα τους εξασφαλίσει μια δουλειά στο μέλλον και θα βελτιώσει και τη ζωή τους γιατί έχουν προοπτικές. Αλλά καμιά φορά αυτό διαρκεί περισσότερο από τέσσερις μήνες και δεν είναι καθόλου εύκολο. Για τις μεταρρυθμίσεις που κάνουν τα κράτη-μέλη Βλέπουμε κατακαιρματισμό της αγοράς εργασίας ε, με ευέλικτες άτυπες μορφές εργασίας με μειωμένο ωράριο για μερικούς νέους μπορεί αυτό να είναι καλό ε, και να τους αρέσει αλλά δεν αρέσει σε όλους και επίσης δεν αρέσει σε εκείνους ε, που θέλουν μόνιμη εργασία είναι ένα νέο ζευγάρι θέλει να ξεκινήσει ε, τη ζωή του, να κάνει οικογένεια, να πάρει δάνειο, στεγαστικό κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται μόνιμη εργασία. Ε, και αυτό χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα παρακολούθηση και όχι από χρόνο σε χρόνο τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει, να αλλάξει ολόκληρη η εργασιακή πολιτική και αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Τώρα μόλι βγαίνουμε από την κρίση, έχουμε περάσει σε ανάπτυξη, θα πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχουν κάποιε εταιρείε που δεν ανοίγουν δουλειέ πλήρους απασχόλησης και μακροχρόνιες και αορίστου χρόνου. Καμιά φορά είναι επισφαλεί μορφέ ευέλικτε με μικρό ωράριο, ε, αλλά δεν είναι πάντα καλής ποιότητας για τους ανθρώπους. Υπάρχει το προσοντολόγιο, skills ε, agenda. Ε, υπάρχουν δουλειές και πάρα πολλές, αλλά και πάρα πολλοί άνεργοι οι οποίοι όμω δεν, αντιστοιχούν με τι ανάγκε τη αγοράς και δεν είναι μόνο νέοι, είναι και μεγαλύτεροι. Και τι διαπιστώνουμε, ότι 40% των εργοδοτών έρχονται και μα λένε ότι εγώ δουλειά έχω, δεν βρίσκω αυτόν που θέλω να προσλάβω, δεν υπάρχουν τα προσόντα. Και γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει αναντιστοιχία των δεξιοτήτων και θα πρέπει να είναι εμβληματική και αυτή η πρωτοβουλία για το, το skill agenda, το θεματολόγιο για τα προσόντα και τι δεξιότητε. σε δέκα σημεία αυτή τη στιγμή όλα εφαρμόζονται εκτός από κάποια βασικά στοιχεία της επαγγελματικής κατάρτισης. Χρειάζεται πιο πολύ δουλειά. Τα άλλα τα έχουμε δρομολογήσει. Και εδώ όμως τι διαπιστώνουμε. Ότι ο κόσμος χρειάζεται κατάρτιση, εκπαίδευση. Ακόμα και όταν στέλνουμε τους νέους στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση, θα πρέπει να είναι εκπαίδευση αυτή αντίστοιχη με τις ανάγκες της αγοράς. Και πολλές φορές που κάνουμε έρευνες και μεταξύ των εργαζομένων σου λένε ότι έχω βρει δουλειά αλλά ε, τα προσόντα μου και οι δεξιότητες είναι πολλαπλάσεις των όσων καλούμε να κάνω στη δουλειά. Άρα και τα προγράμματα σπουδών δεν αντιστοιχούν με τις ανάγκες στην αγορά τις βασικές επίσης γνώσεις και προσόντα και δεξιότητες τις στερούνται πολλοί άνθρωποι. Και στην εκπαίδευση θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και εστίαση ε, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην τεχνική κατάρτιση, στο διτό σύστημα, στην επιχείρηση και στη σχολή. Δεν χρειάζεται να εχεις δυο δύο-τρία πανεπιστημιακά πτυχία. Δουλειά δεν θα βρεις με αυτά τα πτυχία. Χρειάζεται πολύ περισσότερο να δούμε ε, τι κάνουν οι εταιρείε. Έχουμε όλο και περισσότερα προγράμματα και τα κράτη-μέλη αρχίζουν να αλλάζουν οτροπία. Είναι και θέμα ε, κουλτούρας, νοοτροπίας. Αυτή την κουλτούρα που επικρατεί στη Γερμανία και στην Αυστρία δεν μπορούμε να την επιβάλλουμε μέσα σε δύο χρόνια στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Αλλά πρέπει να το καταλάβουν, να κάνουν του μεταρρυθμίσει που χρειάζονται και να προχωρήσουν. Κάνατε μια ερώτηση για τις καθυστερήσεις. Πολλές είναι οι αιτίε. Σας ανέφερα ε, μία από αυτές. Υπάρχει το νησιν χ χρόνια. Ε, διαπιστώσαμε ότι το νησιν 3 οδηγεί σε μια χαλάρωση, έτσι, σε μια διάλυση, ενώ εμείς χρειαζόμαστε πειθαρχία. Ενώ όταν ξεκινάει ένα πρόγραμμα, σου λέει το κράτος μέλος καλά, έχουμε τρία χρόνια μετά τη λήξη που μπορούμε να απορροφήσουμε ε, τα κονδύλια. Αλλά αυτά είναι κονδύλια για να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να τα αξιοποιούν γιατί αλλιώς θα κινδυνεύσουν να τα χάσουν. Το, το νησιν 3 δεν μ' αρέσει. Το, το νησιν 1 δεν, δεν νομίζω. Το νησιν 2 είναι καλύτερο από το νησιν 3. Το, το νησιν 1 νομίζω είναι υπερβολική απέτηση για τα κράτη-μέλη για το PDP μετά το 2020 θα πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό το θέμα οπωσδήποτε. Το ίδιο ισχύει και για την μακροοικονομική ερεσιμότητα, την εξάντε δηλαδή εκ των προτέρων. Το αναφέρετε και εσείς κύριε Σιγητά, θα πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό. Έχουμε δει ότι όλα αυτά που υπάρχουν ως όροι και προϋποθέσεις ε, ευθύνονται για την καθυστέρηση αλλά βοηθούν τα κράτη-μέλη για να απορροφήσουν τα κονδύλια. Άρα αυτά οδήγησαν σε μεταρρυθμίσεις σε κάποια κράτη-μέλη για να μπορούν να απορροφούν αυτά τα κονδύλια και μεταρρυθμίσεις που δεν πιστεύω να γινόντουσαν διαφορετικά. Αλλά θα πρέπει να έχουμε και αυτή την ειλικρίνεια και να το ομολογούμε αυτό. Και να το ξανακοιτάξουμε και για την επόμενη προγραμματική περίοδο μετά το 2020 να κάνουμε προτάσεις και γραπτές. Αλλά τι όρους θα βάλουμε και τι προϋποθέσεις για να μην είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά αυτά και να μην οδηγούν σε καθυστερήσεις. Για τους νέους, τους νέους λοιπόν που βρίσκονται εκτός εργασίας, κατάρτισης, μαθητείας και άσκησης. Το Ταμείο για την καταπολέμηση της παγκοσμιοποίησης και τις μασικές απολύσεις, τι μπορούμε εκεί να κάνουμε. Το Ταμείο αυτό αποδίδει πάντως. 150 εκατομμύρια το χρόνο, αλλά χρειάζονται διάφορες διαδικασίες, χρειάζεται απόφαση του νομοθέτη και είναι μια διαδικασία βαριά και αργή. Την επόμενη προγραμματική περίοδο μήπως να το ε, επιταχύνουμε αυτό από πλευράς διαδικασίας. Το Ταμείο ε, για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση λειτουργεί σε αυτή την περίοδο, κάπου το έχω σημειώσει αυτό. Μια στιγμή να το βρω. Ναι. Όσοι αποφελήθηκαν αυτό το ταμείο, από αυτό το ταμείο απολυμμένοι, ξαναβρίσκουν δουλειά κατά 48%. Αλλά και πάλι με μεγάλες διαφορές ανάλογα με τα προγράμματα μεταξύ των κρατών μελών και στο εσωτερικό των κρατών μελών. Θα πρέπει να δούμε ε, ποιοι είναι οι παράγοντες επιτυχίας για να μπορεί κάποιος να επιστρέψει στην αγορά εργασίας επιτυχώς και να προσαρμόσουμε τα προγράμματα. Επίσης συχνά πρόκειται για μειονεκτούσες περιφέρειες, καθυστερημένες. Δεν είναι εύκολο να απορροφώνται οι άνθρωποι αυτοί και όσοι δεν βρήκαν άμεση δουλειά ή άμεσα δουλειά έχουν τουλάχιστον ε, μία εμψύχωση, έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, έχουν αποκτήσει νέες δεξιότητες έχουν μάθει πώς να ψάχνουν μια καινούργια θέση εργασίας, έχουν δημιουργηθεί μεγαλύτερες ε, εταιρικέ σχέσεις μεταξύ των διαφόρων παραγόντων στην περιοχή των διαφόρων φορέων, ε, δικτύωση, για να μπορεί, γιατί είναι μια ολόκληρη περιφέρεια. 150 εκατομμύρια το χρόνο, δεν απορροφώνται όλα, ίσως επειδή είναι πολύ μεγάλη η ε, διαδικασία και πολύ βαριά και μέχρι να κινητοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της. Στο μέλλον όμως θα πρέπει να αυξηθεί αυτό το ποσό γιατί περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερα δεινά με την παγκοσμιοποίηση και την ψηφιοποίηση και θα πρέπει να έχουμε ένα, ένα buffer, ένα, ένα μαξιλαράκι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την οικονομία μας να το αντιμετωπίσει. Να δούμε τι λέει η δική μας νομοθεσία για την αναθεώρηση και τις μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι πάντα εύκολο. για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, ε, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Η νομοθεσία μας λέει ότι θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων τα συνδικάτα, εργαζόμενοι ενώσεις κτλ. Ε, θα λάβουμε μία έκθεση προσεχώς για το πώς τα χειρίζονται αυτά τα κράτη-μέλη και πώς τα εφαρμόζουν στην πράξη οι επιχειρήσεις για να δούμε πώς χρειαστούν περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες. Οι επιλογές ε, απλούστευσης κόστους, simplified cost options, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και αυτό είναι θετικό. Μόλις 7% των ε, πληρωμών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου γίνονταν με αυτό το σύστημα. Τώρα έχουμε φτάσει στο 35%. Εφτά κράτη-μέλη έχουν ξεπεράσει το 50%, το είπα και εισαγωγικά, και προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε. Ποια είναι τα προβλήματα, για ποιο λόγο διστάζουν καμιά φορά τα κράτη-μέλη. Είναι η άγνοια ότι όταν δεν ξέρεις ένα σύστημα δεν το προτιμάς, δεν το χρησιμοποιείς, το φοβάσαι. Και τα κράτη-μέλη πραγματικά φοβούνται αυτή την ανασφάλεια δικαίου. Γιατί εμείς το προωθούμε γιατί σε αυτή την περίοδο και αυτό ενισχύει την ασφάλεια δικαίου. Μπορούμε να δουλέψουμε με κατεξοδότηση πράξη για τα κράτη-μέλη. Εκ των προτέρων να έχουμε ορίσει πώς θα γίνει αυτό. Και ήδη είναι 14 τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και είναι 7 δισεκατομμύρια η συνολική δαπάνη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Κάνουμε και πακέτα έτοιμα προς χρήση για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και τα κρατημέλη και οι ενδιαφερόμενοι και οι δικαιούχοι να μην στείνεται ένα πρόγραμμα από την αρχή ενέργου μπορούν ε, να πάρουν μια έτοιμη προκάτληση. Και στο Omnibus το προτείνουμε. Θέλουμε να φτάσουμε προς το 50%. Μήπως να αυξηθεί το κατόφλι 100.000 ευρώ, όχι 50.000 ευρώ που είναι σήμερα για να χρησιμοποιείται αυτή η νέα διαδικασία. Θα βοηθήσει και αυτό. Και επίσης να χρησιμοποιήσουμε νέες μορφές χρηματοδότησης. Να έχουμε ένα στόχο εκ των προτέρων, να στείλουμε ένα έργο και όταν φτάνει κάποιος στον επιθυμητό στόχο να παίρνει και τα ποσά αυτά χωρίς κάθε φορά να πρέπει να δικαιολογεί την κάθε απόδειξη και το κάθε τιμολόγιο. Αυτό είναι νέος τρόπος χρηματοδότησης που μπορεί να εθαρρύνει τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν με την απλοποιημένη διαδικασία για τις μικροπιστώσεις, μικροδάνεια που χορηγούμε και συμμετέχουμε, αλλά και δάνεια και εγγυήσεις. Έχουν εξαντληθεί τα κονδύλια που προβλέπονται. Είναι ελκυστικός αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης και χρησιμοποιείται με καλό ε, τρόπο. Γι' αυτό ζητήσαμε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ των διαφόρων τύπων και μορφών ε, που χρηματοδοτεί το EASY. Ε, Προφανώ πάντα έχει κάποιον ενδιάμεσο και ο ενδιάμεσο πληρώνεται για την υπηρεσία που σου παρέχει. Λέτε για τι τράπεζε και τι προμήθειε. Μπορεί να δούμε πώ θα βελτιωθεί στο μέλλον. Εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων που έχει τριπλό α και θέλουμε να το διατηρήσουμε. Και αυτοί που είναι τόσο αξιόπιστοι πιστοτικά ιδρύματα έχουν και μεγάλο κόστος για τα, τις μικροπιστώσεις αυτές, τα πολύ μικρά δάνεια. Αυτό που με ενδιαφέρει, αυτό που με ανησυχεί είναι ότι αυξάνεται η αγορά. Πολλές φορές ε, οι άνθρωποι αυτοί που παίρνουν αυτό το μικρό δάνειο ε, είναι αυτοποσχολούμενοι. Δημιουργούν επιχειρήσει με βιώσιμες ε, θέσει εργασία και προσλαμβάνουν και κόσμο μετά και μπορούμε να δημιουργήσουμε 150 και 170 χιλιάδες θέσεις εργασίας με μια νεοφυή εταιρεία. Αυτό που θέλουμε είναι να αυξηθεί η αγορά η βάση των ανθρώπων. που ε, προσφεύγουν σε αυτά τα δάνεια. Και θα πρέπει να έρθουν πιο κοντά οι τράπεζες και το επίσημο τραπεζικό σύστημα με την κοινωνική οικονομία και ε, ε να μάθουν περισσότερο τι σημαίνει κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και αντίστροφα ε, για να μάθουν και εκείνοι πώς δουλεύουν οι τράπεζες και τι γίνεται με τις επιδοτήσεις, με τα δάνεια και τις εγγυήσεις. Αυτά. Α, και άλλη μια ερώτηση που κάνατε για την αρχιτεκτονική του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου δεν το κατάλαβα. Ίσως διμερώς να το ξανασυζητήσουμε ή κάποια στιγμή αργότερα. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας με τρόπο ικανοποιητικό. Αλλιώς ξαναρωτήστε με. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Επιτροπή. Πολλές ερωτήσεις, πολλές και απαντήσεις. Τώρα θα απευθυνθώ στους κοιότητες ηγητές. Η κυρία Γιαλασέντερ καταρχήν. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στον κύριο Πυρίνσκι που είναι στην Επιτροπή Απασχόλησης. Θα το δώσετε μετά φαντάζομαι το λόγο. Καλωσορίζω την Επίτροπο κυρία Τάισεν. Ο κύριος Τσέλερ ήταν ε, εξαντλητικός, ε, λίγο, λίγα μένουν να πω εγώ. Όμως έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι εμεί εμείς εξετάζουμε την ε, χρήση των κονδυλίων και τα προγράμματα εφαρμής του κοινωνικού ταμείου, την, ε, τα προγράμματα εγγύσεων ε, για τους νέους, αλλά και τις υποτροφίες και άλλα προγράμματα με αρκετά υψηλά κονδύλια του προγράμματος Οριζοντας 2020. Είναι ένα πρόγραμμα για την καινοτομία, όπως γνωρίζετε, που έχει δύο σημαντικές πτυχές, δύο σημαντικούς πυλώνες. Πρώτον, τις ενισχύσεις που δίνονται σε ομάδες ερευνητών, ε, που εργάζονται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτές τις ενισχύσεις είναι υπό τη μορφή υποτροφιών σε σπουδαστές και από την άλλη μεριά ένα άλλο μεγάλο κομμάτι σε ερευνητικές ομάδες ε, με συμβάσεις ε, σε που συνάπτονται με καθηγητές, επιστήμονες κλπ Όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Έχουμε αντιληφθεί τελευταία το εξής. Είτε οι δικαιούχοι είναι κυβερνήσεις, είτε είναι, είτε είναι οι τελικοί δικαιούχοι, οι σπουδαστές και οι καθηγητές, οι ερευνητές, τα ερευνητικά κέντρα κλπ. Έχουμε συμπεράνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο τύπους πρόσβασης, σε δύο τύπους ε, ε, απασχόλησης. Απ' τη μία μεριά υποτροφίες σε σπουδαστές και συμβάσεις ε, για ε, επιστήμονες και από την άλλη μεριά το κοινωνικό ταμείο που παρέχει βοήθεια, ενίσχυση ε, για την πρώτη απασχόληση και για την κατάρτιση. Και οι προσεγγίσεις αυτές είναι διαφορετικές. Δεν είναι ομογενής η κατάσταση. Ε, η ιστορική αδράνεια του κοινωνικού ταμείου έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές οι νέοι, οι νέοι που δεν βρίσκονται σε εκπαίδευση κατά τη εργασία ε, έχουν την εντύπωση, τους δημιουργείται η εντύπωση ότι ε, δεν είναι καλή υποψήφοι για επιχειρήσεις ή για ενδεχόμενους εργαζόμενους. Αντίθετα, στο πλαίσιο του ορίζοντας 2020, παρόλο ότι ε, δεν είναι πολύ ψηλότερα τα ποσά των υποτροφιών εκεί, έτσι, δεν είναι τίποτα τεράστια ποσά, παρόλα αυτά, οι υποτροφίες που δίνονται μέσω του 2020 ε, εξαιτία του, του φορμάτ που έχουν ε, του δημιουργούν την εντύπωση ότι οι δικαιούχοι είναι εξαίρετοι υποψήφοι για εργασία. Και εν πάση περιπτώσει ότι οι ίδιοι θεωρούν πως είναι πιο απασχολήσιμοι επειδή έλαβαν μια υποτροφία του ορίζοντα 2020. Από την άλλη μεριά, οι ενισχύσει του κοινωνικού ταμείου δεν θεωρούνται εξίσου καλέ. Δεν θεωρούν οι ίδιοι δικαιούχοι ότι τους βοηθούν εξίσου. Ζητήσαμε μια συγκριτική μελέτη και θα ήθελα να ρωτήσω και εσάς. Με τον κύριο Μουέδας έχετε συζητήσει την δυνατότητα να ανταλλάξετε τις βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε όλες οι ενισχύσεις, όλα αυτά τα τεράστια ποσά τα οποία ε, δαπανώνται να ε, οδηγούν προς την αριστεία χωρίς διαφορές ανάμεσα στους διαφορετικούς τύπους βοήθειας. Μήπως θα μπορούσε ο ένας να μάθει από τις καλές πρακτικές του άλλου. Και μετά, κάτι για το μέλλον. Είναι πολύ θετικό το ότι οι, τα τρία ε, όργανα έθεσαν, θέτ, άρχισαν να θέτουν σε εφαρμογή τον κοινωνικό πυλώνα. Είναι ένα είναι μια εξέλιξη πολύ αισιόδοξη. Γιατί αυτός ο πυλώνας μπορεί να ε, στηρίξει όλες αυτές τις φιλοδοξίες περί κοινωνικής δικαιοσύνης κλπ. Ποια είναι η άποψή σα για τις ε, συστάσεις μας στην απαλλαγή του 2016 σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό πυλώνα και τα δύο προγράμματα τα οποία τον στηρίζουν και βέβαια ενδεχομένω και άλλες πρωτοβουλίες. Πιστεύετε ότι θα είναι αρκετά για να στηρίξουν αυτόν τον κοινωνικό πυλώνα στο μέλλον. Ποια θα διατηρούσατε και ποια θα αλλάζατε. Είμαι και ως συγγήτρια για, την, ε, για τους φιλελεύθερους, οπότε έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να περιορίσω ε, τον, την παρέμβασή μου σε θέματα δημοσιονομικού ελέγχου, ελέγχου του προπολογισμού ε, και να μην επεκταθώ σε θέματα απασχόλησης, γιατί αλλιώς θα μου πάρει πάρα πολύ ώρα. Καταρχήν συμφωνώ με τον κύριο Τσέλερ σε ό,τι αφορά τις περίπλοκες διοικητικές δομές και εγώ θέλω να το υπογραμμίσω. Αυτή η περιπλοκότητα δυσχεραίνει τη δουλειά των δικαιούχων. Βλέπω ότι η απλοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει και έχει θετικά αποτελέσματα. Τα simplified cost options ε, μειώνουν ενδεχομένως το διοικητικό άχθος των δικαιούχων και προφανώς και τον κίνδυνο λάθους. Αλλά η ερώτηση είναι γιατί χρειάζεται να τις προωθήσουμε και να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να τις χρησιμοποιούν εφόσον γνωρίζουν ήδη το όφελος. Γιατί τα κράτη-μέλη ε, δυσκολεύονται, ε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό. Και μετά, κρατικές ενισχύσεις. Πολλά κράτη-μέρη μου λένε ότι η περιπλοκότητα των κανόνων είναι θέμα. Κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιεί διαφορετικούς ορισμούς. Ε, ιδιαίτερα το θέμα του ανταγωνισμού στις παραμεθόρεις περιοχές. Ε, αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Το υπερπλοκότητα των κανόνων κρατικής σχέσης ε, σχεδόν είναι απαγορευτική για να προκειμένου να δοθούν ε, δωρεάν ενισχύσεις, επιδοτήσεις δηλαδή, σε αυτούς που πιο πολύ τις χρειάζονται. Αυτά. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πυρίνσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ όσο πιο σύντομο γίνεται. Ε, περιμένω λίγο την κυρία Τάισιν και τον Σερβόση να τελειώσουν αυτά που λένε. Ευχαριστώ, Επίτροπε που είστε εδώ σήμερα. Τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη έχει σχέση με αυτό που ήδη μιλήσαμε, ε, για αυτό που ήδη είπαμε, για την απροφητικότητα του 5,1% για το κοινωνικό ταμείο. Και αναφέρατε τρεις λόγους. Ε, ο ένας λόγος είχε σχέση με το νησιντρία ε, Δεύτερον, οι εξάντε ερεσιμότητας, ερεσιμότητες όπως απαντήσατε στην ερώτηση 17 και ένα τρίτο λόγο ε, που αναφέρεται στη γραπτή σας απάντηση ότι τα κράτη-μέλη είναι πολύ προσεκτικά εξαιτία των ετήσιων λογαριασμών που έχουν εισαχθεί και του κινδύνου για δημο... και δημοσιονομικές διορθώσεις. Πιστεύετε ότι αυτός ο λόγος πρέπει να ε, αυτό το, αυτή η κατάσταση πρέπει να διορθωθεί και πώς. Ε, και άλλες δύο ερωτήσεις για το Κοινωνικό Ταμείο και την πρωτοβουλία για τους νέους. Ε, οι διαχειριστικές αρχές που έχουν οριστεί πλέον μπορούν να, μπορεί η θητεία τους ε, να ανανεωθεί και για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις εμπειρίες των κρατών μελών, όπως είπατε, σε μερικές περιπτώσεις οι κρατικές αρχές πολύ, ε, έρχονταν σε επαφή με μη κυβερνητικέ κυβερνητικού οργανισμού όπω τα συνδικάτα, ενώ σε άλλε χώρε δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ε, έχει αυτό, δίνει αυτό διαφορετικά αποτέλεσματα στην απορροφητικότητα. Κατόπιν, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ερώτηση 2. Στην ερώτησή μας αναφερόμασταν στην προσμονή η Επιτροπή να λάβει την αξιολόγηση σε χώρα και για τις κοινωνικές πτυχές του εξαμήνου. Εσείς λέτε στην απάντησή σας ότι η αυτή η αξιολόγηση ε, είναι ένα έργο όλης της Κομισιόν και όχι μόνο της Γενική σας Γενικής Γραμματείας. Τι, Γενικής Διεύθυνσης, Όμως, με τον κοινωνικό πυλώνα έχουμε, έχουν δημιουργηθεί υψηλότερε απαιτήσει. Ίσως θα έπρεπε να δούμε με πολύ περισσότερη προσοχή λοιπόν αυτές τις κοινωνικές πτυχές και αυτό με φέρνει στην ε, ερώτηση 7 για τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων στο τμήμα τη Οικονομικής και Νομισματική Ένωσης. Λέτε όμως, σε ό,τι αφορά την πρώτη σύσταση, ε, ότι αυτή αφορά μόνο την ζώνη του ευρώ και έχει σχέση με την Δημοσιονομική και Οικονομική Ένωση την ε, διακυβέρνηση και τη λογοδοσία. Η τελευταία σας φράση λέτε ότι στην αρχιτεκτονική θα πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα για μεταρρυθμίσεις και ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ΟΝΕ θα, εξασφα... θα πετύχει τους αρχικού της στόχους για περισσότερη απασχόληση και οικονομική και κοινωνική συνοχή. Στην με δεδομένο ότι τώρα αρχίζουμε να εφαρμόζουμε τον κοινωνικό πυλώνα, πιστεύετε, δεν πιστεύετε ότι θα οδηγηθούμε σε μεγαλύτερη σε διαφορά μεταξύ της ζώνης του ευρώ και των υπόλοιπων χωρών. Δεν πιστεύετε ότι θα αποκλίνουν αυτές οι δύο ζώνες. Έχω την εντύπωση ότι θα κινηθούμε αντίθετα από την κατεύθυνση τη κοινωνική συνοχή. Πρόεδρο, ευχαριστώ κύριε Πυρινσκή. Κύριε Τίσεν, ελπίζω ότι προλάβατε να σημειώσετε όλε τι ερωτήσει. Ήταν αρκετέ. Μία μου ξέφυγε, αλλά θα μου την πούν οι συναδελφοί μου, οι βοηθοί μου disait dans notre question 2. Mm C'est Uh, May I maybe ask first the Court of Auditors because maybe... Μήπως δώσω το λόγο στο Ελεκτικό Συνέδριο πρώτα. Χρειάζεται... Εντάξει, εσείς, οκ. Okay. Για την κυρία Γιάλα Σέντερ. Συγγνώμη, θα το πω Ολλανδικά. Ε, Ορίζον 2020 και τα δικά μας κονδύλια και τα μία. Είναι πολύ καλή ανάλυση για αυτό που άκουσα ότι όταν ε, έχουν μια δουλειά ε, οι άνθρωποι ε, αισθάνονται ότι είναι πολύ ε, καλό αυτό που κάνουν, ότι μπορούν να προχωρήσουν, ότι υπάρχει μια αναγνώριση και μόνο από το γεγονός ότι έχουν επιλεγεί. Ε, τώρα για το ποιος είναι δικαιούχος για τα ε, κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή άλλων ταμείων που είναι στις δικές μας αρμοδιότητες, ότι δεν είναι πάντα τόσο ελκυστικά ότι ορίζον 2020 και τα κονδύλια ας πούμε, προς την έρευνα για της αριστείας είναι πιο ελκυστικά, είναι πιο ε, Άμεση απασχόληση ο κόσμος βρίσκει καλύτερη και πιο γρήγορα δουλειά από το επίπεδο αριστείας ε, στον ορίζοντα 2020 και τα δικά μας κονδύλια δεν είναι τόσο ε, θεαματικά τα αποτελέσματα, τόσο συναρπαστικά ή τόσο γρήγορα. Αλλά ορίζοντα 2020 ακριβώς έχει σχέση με την αριστεία και με την έρευνα. Δηλαδή αυτό βοηθάει τους ανθρώπους που έτσι κι αλλιώς έχουν καλές προοπτικές, είναι ερευνητές υψηλού επίπεδου που θα βρουν δουλειά έτσι κι αλλιώς. Ενώ το ESF, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν δυσκολίες να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία, που δεν τα πήγαν τόσο καλά στο σχολείο, που χρειάζονται μετεκπαίδευση, που βρίσκονται κάπου στη μέση, αλλά χρειάζονται μια ενθάρρυνση για να βγουν από την κρίση που γνώρισαν, να επανέλθουν στην αγορά εργασία και στην κοινωνία στα καλύτερα του χρόνια και να λειτουργήσει και στην οικονομία. Είναι διαφορετική η στόχη λοιπόν της χρηματοδότησης και οι ομάδες στόχοι επίσης. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να ε, βοηθήσουμε τους ανθρώπους να πιάνουν τόπο τα χρήματα. Και οι άνθρωποι αυτοί να γνωρίζουν επίση το σεβασμό των υπόλοιπων. Σας παραπέμπω στην περασμένη εβδομάδα που είχαμε ε, την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Επαγγελματική Κατάρτιση, Εκπαίδευση και Δεξιότητες και ήμουν όλη τη βδομάδα σε διάφορες δραστηριότητες ανά τις Βρυξέλλες και πρέπει να σας πω ότι εκείνοι που συμμετείχαν, που ήρθαν να δώσουν τη μαρτυρία τους στη δική τους προσωπική ε, ιστορία εποφελήθηκαν πάρα πολύ χάρη στα δικά μας ε, μέσα. Και την περασμένη φορά το ακούσαμε που ήταν η πρώτη φορά που διοργανώσαμε αυτή την εβδομάδα ότι πόσο βοήθησε στη χώρα τους, στην περιοχή τους κτλ. Ε, αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και αυτό είναι στην ατζέντα, στο θεματολόγιο ε, των δεξιοτήτων, οι άνθρωποι που παρακολουθούν τη τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να χαίρουν μεγαλύτερη εκτίμηση στην κοινωνία, να είναι καλή η εκπαίδευση, να είναι ελκυστική και αυτό έχει να κάνει και με την ποιότητα τη ίδια ε, της εκπαίδευσης αλλά και πόσο βλέπουν στην κοινωνία, πώς αξιολογείται αυτό ο άνθρωπο μετά και πού κατατάσσεται. Αύριο με τον συνάδελφο Μοέδας ε, θα πάμε στη Λισαβόνα σε μία ε, διάσκεψη. Αυτή έρχεται σήμερα βέβαια, αλλά επειδή εγώ έπρεπε να βρίσκομαι εδώ, θα πάω το βράδυ αμέσω μετά. Για την κοινωνική καινοτομία λοιπόν, μαζί με τον συνάδελφο Μοέδα, που είναι αρμόδιο για τον ορίζοντα 2020, συμμετέχει και το κοινωνικό ταμείο και είναι πάρα πολύ καλό και για μένα μεγάλη ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει για το μέλλον. Πραγματικά στενίζω τα όσα λέτε και τη συστασία σα και θα το συζητήσω με τον συνάδελφο Μοέδας στη Λισαβόνα. Τι άλλο με ρωτήσατε. Ο συνάδελφος Πυρίνσκι. Ε, τα στοιχεία για την απορροφητικότητα. Είναι χαμηλή η απορροφητικότητα με διάφορα στοιχεία. Ευτυχώς τώρα καλύπτουμε αυτή τη διαφορά. Νήσιν 3, εξάντε ρεσιμότητα. Ο κίνδυνος να έρθουν οικονομικές διορθώσεις και να επιστραφούν ε, δισεκατομμύρια. Ε, αυτό έχει να κάνει και με τις καθυστερήσεις. Γι' αυτό υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις, ότι περιμένουν να βεβαιωθούμε όταν ε, ζητάμε ανάκτηση των πόρων, όταν κάνουμε μια τέτοια αξία, για να μην χρειαστούμε διορθώσεις. Αυτές γίνονται όταν δεν έχει εντοπίσει το κράτος μέλος το ίδιο το σφάλμα ε, όταν αξιώνουν κάποιες πληρωμές οι δικαιούχοι. Αυτό είναι πραγματικά ένας ε, παράγων καθυστέρησης, αλλά το όφελος είναι μεγαλύτερο από το κόστος. Καλύτερα να βεβαιωθούν τα κράτη-μέλη ότι τα έχουν κάνει όλα καλά και ας καθυστερήσουν λίγο. Εμείς βασιζόμαστε στα αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων που κάνουν τα κράτη-μέλη για να μην πολλαπλασιάζουμε τους ελέγχους και τελικά να βάζουμε μόνο λεφτά σε λογιστικούς ελέγχους και συλλογή στατιστικών στοιχείων. Γι' αυτό ε, τα χρήματα δεν θα πρέπει να σκορπίζονται δεξιά και αριστερά, αλλά σκοπός τον οποίο διατίθενται. Για μας είναι μεγαλύτερος ο παράγοντας αξιοπιστίας να περιμένουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν τους ελέγχους τους, να μας στείλουν επίσημα στοιχεία και μετά να προχωρήσουμε. Έχει βελτιωθεί το αποτέλεσμα ή βελτιώνεται όταν, στην απορρόφηση ε, όταν υπάρχει καλύτερη συνεργασία των κρατών μελών με τις ΜΚΟ και τα συνδικάτα. Δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν έχω τέτοια στοιχεία. Μπορεί, έχετε εσείς τέτοια στοιχεία. Υπάρχουν χώρες όπου υπάρχει ένας καλός κοινωνικός διάλογος και όπου οι κοινωνικοί εταίροι συνεργάζονται άγαστα με τις ε, κρατικές αρχές. Είναι καλύτερα και τα κοινωνικά αποτελέσματα. Όταν υπάρχει καλή συνεννόηση και συνεργασία μπορεί να βοηθήσει και όλα βελτιώνονται. Μπορεί και η απορρόφηση των πόρων, αλλά δεν έχουμε τέτοια στατιστικά στοιχεία. Όταν τα πάρουμε, τα πάρουμε θα σας τα διαβιβάσω. Τι άλλο με ρωτήσατε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τον κοινωνικό πυλώνα. Οι συστάσεις στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αναχώρα προκύπτουν από συνεννοήσεις μεταξύ διαφόρων γενικών διευθύνσεων. Και εμείς πιέζουμε πάρα πολύ για τα κοινωνικά, θα το φαντάζεστε. Το από την παρούσα θητεία, μου είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ, φρόντισε το ευρωπαϊκό εξάμεινο να γίνει πιο κοινωνικό, να υπάρξουν εξέχοντα κοινωνικά στοιχεία. Κάνουμε τη δουλειά μας. Το βλέπω στις συστάσεις αναχώρα και στην ετήσια έκθεση για την ε, ανάπτυξη και σε όλη την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου υπάρχει μια κοινωνική απόχρωση πιο έντονη. Έχουμε μια σειρά δικτών, κοινωνικών δικτών που έχουμε συμπεριλάβει όλους από την αρχή ε, στη νέα άσκηση του εξαμήνου που λανσάραμε την περασμένη εβδομάδα και θα φανεί πραγματικά ότι έχουμε κάνει πολλή δουλειά για τον πυλώνα. Τώρα, τι προέρχεται στο, στο εξάμεινο από την Τάισεν, από το Μοσκοβισί από τον Ντομπρόφσκης, δεν θα το γράφει τόσο ρητά η κάθε σύσταση αναχώρα. Ε, από κοινού γίνεται η προσπάθεια, αλληλοεμπνεόμαστε, συνεργαζόμαστε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσει και ο κοινωνικός πυλώνας. Δεν περιμένετε και τίποτα λιγότερο από εμάς ε, ο ναι, εμβάθυνση τη οικονομική και Νομισματικής Ένωσης. 6 Δεκεμβρίου θα έρθει αυτή η δέσμη μέτρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώ θα έχει νέα αυτή η αρχιτεκτονική. Δεν μπορώ να το πω ακόμα γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Πάντω πιστεύουμε ότι στην Ευρωζώνη που έχουμε το ίδιο νόμισμα και λιγότερα εργαλεία προσαρμογής όταν υπάρχει μια συμμετρία, δηλαδή δεν μπορούμε ο καθένας ξεχωριστά να κάνει υποτίμηση του νομίσματος. Είμαστε στο ίδιο σύστημα και σε ίδια πολιτική νομισματικά. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίζουμε η συνοχή να είναι πιο ισχυρή ε, από ό,τι στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν είναι ότι το θέλουμε, το οφείλουμε. Αλλά ανέκαθεν το είπαμε από τη στιγμή της σύλληψης του κοινωνικού πυρόλα ότι θα πρέπει να ισχύει και για την ε, Ευρωζώνη, αλλά καλύτερα για όλους. Και χαίρομαι που αυτό επικράτησε για όλους, 28 και προσεχώς 27. Ε, όλοι κάνουμε κοινωνική πολιτική και η συνοχή πρέπει να παραμείνει ε, και να αυξηθεί και στους 27 και τελικά όλοι θα γίνουν μέλη της Ευρωζώνης με μια εξαίρεση τη Δανία. Αν δούμε όμως πώς εξελίσσεται και πώς εμβαθύνεται ε, ο ναι, θα πρέπει να βρούμε ένα μαξιλαράκι, ένα buffer, όταν έχουμε ασύμετρους ε, κραδασμούς, ε, κάπως να υπάρχει μια ταχύτερη αντιμετώπιση. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα χρησιμοποιηθεί, πώς θα χρηματοδοτηθεί, δεν ξέρω, θα το δούμε. Όλα αυτά στα πλαίσια του εξαμήνου. Ξέρετε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Μέλη της Ευρωζώνης και μη για τα μέλη της Ευρωζώνης μπορούμε να επιβάλλουμε και πρόστιμα και κυρώσεις όταν δεν σέβονται το σύμφωνο σταθερότητας. Οι υπόλοιποι δεν έχουν κανένα σύμφωνο σταθερότητας να σεβαστούν, αλλά η συνοχή πρέπει να ισχύει για όλους. Τι άλλο έχω. Κρατικές ενισχύσεις. Σύντομα, σύντομα. Ε, και για κρατικέ κρατικές έγινε μια ερώτηση. Νομίζω ότι θα πρέπει κυρίως να κοιτάξουμε ε, τις διαδικασίες. Είπατε κι εσεί ότι είναι πολύ βαριέ και μήπω να κοιτάξουμε τους κανόνε de και για τα τέτοια έργα να μην γίνονται εξαιρέσει. Γιατί η διαδικασία κρατικών ενισχύσεων είναι πραγματικά μια βαριά διαδικασία. Και στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να δούμε πώς μπορούμε να προβλέψουμε αυτή τη ρύθμιση. Οι απλουστευμένες επιλογές κόστους. Γιατί δεν είναι τόσο ολικιστικές για τα κράτη-μέλη όπως είχαμε φανταστεί. Μα δεν το γνωρίζουν αυτό τα κράτη-μέλη. Είναι κάτι το καινούριο ή εκείνοι που χειρίζονται τα έργα. Και ε, όταν κάτι δεν το γνωρίζεις δεν το αγαπάς κιόλας όπως λέει μια Ολλανδική παροιμία. Αλλά είναι πιο εύκολο ε, να έχουμε στάνταρ διαδικασίες παρά να πρέπει να δικαιολογούμε μέχρι την τελευταία απόδειξη. Αυτά. Μπορείτε να απαντήσετε μερικές ερωτήσει και γραπτός αν θέλετε. Η κυρία Βάνοβα από το ελεγκτικό συνέδριο γιατί νομίζω ότι έχει και ίδια να απαντήσει μια ερώτηση. Και μετά στον κύριο Τσέλερ για να κλείσει. Κύριε Βάνουμα. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Ο εισηγητής έθιξε σημαντικά ζητήματα και την ε, μείωση του ποσοστού λάθους αλλά και την ε, αύξηση της επίδοσης. Της απασχόλησης, συγγνώμη. Ε, η απασχόληση αυξήθηκε, ωραία, αλλά σίγουρα έχουν βελτιωθεί οι μακροοικονομικές συνθήκες συνολικά. Και αυτό είναι ένα βασικό ρόλο. Ε, λόγος. Αυτή, αυτό ήταν και ένα από τα συμπεράσματα ε, της σύσκεψης για την απασχόληση που έλαβε χώρα εδώ στο Κοινοβούλιο. Ότι η απασχόληση των νέων και η εγγύηση της απασχόλησης των νέων χρειάζονται μια συνολική απάντηση, ολιστική. Μετά μιλήσατε για τις νέες προκλήσεις κοινωνικής πολιτικής και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτήν την ευκαιρία να σας πω ότι το 2018 θα ετοιμάσουμε ένα briefing paper, ένα ενημερωτικό έγγραφο για την ένταξη, ενσωμάτωση των προσφύγων, των μεταναστών. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό ε, έχουμε κάποια αριθμητικά στοιχεία τα οποία δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά. Το 48% των νέων ε, παραμένουν στα μέτρα έξι μήνες αφότου έλαβαν την ενίσχυση. Αυτό ε, είναι ο συνολικός μέσος από την αρχή. Η μέτρηση όμως της βιωσιμότητας χρειάζεται χρόνο. Ίσως τα αποτελέσματα θα, θα ήταν διαφορετικά αν μετρούσαμε τώρα μόνο. Τώρα για την ερώτηση 25 που αφορούσε την Κομισιόν να σχολιάσω και εγώ γιατί η ερώτηση σχετίζεται με τις αδυναμίες που εντόπισε το ελεκτικό συνέδριο παράδειγμα η έλλειψη σαφήνες στρατηγικές με συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα, ε, έλλειψη αξιολόγηση χρηματοδότηση, ε, έλλειψη επανεπαρκής ενσωμάτωση, το είπατε και εσείς κυρία Επιτροπέ. Κανένα από τα κρατημέλη τα οποία επισκεφθήκαμε δεν έχει ολοκληρώσει την ανάλυση ε, μη καταλληλότητα των προσόντων. Μόνο η Ιρλανδία. Της μια ε, μη αντιστήχησης προσόντων. Ναι. Η Κομισιόν το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να καλέσει τα κράτη-μέλη, να κάνει εκκλήσεις, αλλά τελικά τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν αυτές τις στρατηγικές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, απλοποιημένες ε, επιλογές κόστους. Θα επαναλάβω αυτά που είπα την περασμένη εβδομάδα από τις 135 ε, συναλλαγές ε, του περασμένου έτους δεν εντοπίσαμε κανένα λάθος κανένα μετρήσιμο λάθος τώρα εκ εκτός από την ενημερω... το ενημερωτικό έγγραφο για την απλοποίηση ε, θα ετοιμάσουμε και άλλο υλικό, πιο τομεακό για παράδειγμα για τη γεωργία σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες απλοποίησης. Συμφωνώ με την Κομισιόν, χρειάζεται χρόνο. Θα πρέπει τα... οι δικαιούχοι να μάθουν τις διαδικασίες και ελπίζω ότι ε, τα έγγραφα τα οποία θα παρουσιάσουμε του χρόνου θα σας διαφωτίσουν περισσότερο. Αυτά. Uh, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ιβάνοβα και ο κύριος Ζέλερ της ε, τελευταίες του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Ιβάνοβα και την κυρία Τάισεν για τις ε, παρεμβάσεις τους. Για το θέμα της αρχιτεκτονικής των οικονομικών, ίσως εγώ δεν μην ήμουν αρκετά σαφής. Ε, τι ερωτούσα; Έχουμε πάρα πολλές πηγές χρηματοδότησης από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον ESM για χώρες ε, χρεωμένες στο ευρώ, ο μηχανισμός σταθερότητας. Ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζει 60 δις δάνεια κάθε χρόνο. Άλλες πηγές, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Επίσης έχουμε και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και σχέδιο Juncker ε, γνωστό και ο σχέδιο Juncker και εκτός από τον Ευρωπαϊκό Προεπολογισμό τα διαρθωτικά ταμεία, εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και μετά με διάφορα καταπιστεύματα που τα διαχειρίζεται κάποιος εξωτερικά, ε, ε, αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η ζωή εκείνων που ελέγχουν τον προπολογισμό από τη μια και από την άλλη σε όλο αυτό το γαλαξία και τον εφέλωμα ε, ε, διερωτώ με τι ρόλο παίζουν τα διαρθρωτικά ταμεία ε, που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό άμεσα και ποιο είναι το μέλλον τους. Πριν από λίγα χρόνια μας είχαν πει ότι το κατεξοχή εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσων για να δημιουργήσει Θέση εργασίας και ανάξη είναι τα διορθωτικά ταμεία. Αυτό περίπου δεν αναφέρεται πια από κανέναν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν πρόκειται για την ανάπτυξη και την απασχόληση και την ε, ενίσχυσή τους οικονομικά από το ίδιο μου το παρελθόν και την προηγούμενη εμπειρία μου γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 η ανεργία στη Γερμανία ήταν τελείως διαφορετική από τη σημερινή ευνοϊκή κατάσταση. Στην πατρίδα μου στο Βερολίνο ήταν πάνω από 25% η ανεργία των νέων και 20% του συνολικού πληθυσμού. Και το καταφέραμε να το ξεπεράσουμε μόνο επειδή είχαμε ευρωπαϊκά κονδύλια και του Κοινωνικού Ταμείου. Από την άλλη, Γνωρίζω ότι για να υλοποιηθούν όλα αυτά χρειάζονται περίφημες δομές για τη διάρθρωση εξού και Αν δεν είναι δεδομένη αυτή, που δίνουν στο νέο τέσσερις μήνες απασχόληση και μετά τον, τον αφήνουν πάλι εκτεθειμένο στο δρόμο ή τον καταρτίζουν για ένα επάγγελμα που δεν έχει καμία επαγγελματική προοπτική. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη συνδιαλλαγή για τον προπολογισμό και το 2018 θέλει να ε, ενισχύσουμε ε, τα μέσα για την ευρωπαϊκή ε, εγγύηση για την νεολαία και υποτίθεται ότι ο Ισπανός και ο Πορτογάλος πρέσβης είπαν ε, φήμη είναι αυτή ότι δεν χρειάζεται να αυξηθεί η πυρκοδότηση γιατί είναι πολύ δύσκολα στην απορρόφηση αυτά τα κονδύλια. Και μετά αυτή η φήμη εξαφανίστηκε και πάλι. Δηλαδή πραγματικά αυτή η σέμα για να πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα, αλλά δεν είναι το παν πάντα το χρήμα. Κάτι άλλο που είχα ρωτήσει, δεν άκουσα να απαντήσατε, μπορεί να απαντήσατε, για τα 200 εκατομμύρια που ανακτάται από την Ισπανία και την ε, Ιταλία από την περίοδο 2000-2006. Γιατί χρειάστηκαν 10 χρόνια μέχρι να γίνει αυτή η επιστροφή. Δεν άκουσα να απαντήσατε. Μπορεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία στην κοινωνική πολιτική και στο μέλλον. Thank you very much, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζέλερ. Επίτροπε. Θέλετε σύντομα να επανέλθετε σε αυτό το τελευταίο ερώτημα που δεν απαντήθηκε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Σεγητά. Ναι, για την τελευταία ερώτηση. Γιατί χρειάστηκε μια δεκαετία για τα χρήματα για την Ιταλία. Αυτό είναι θέμα στο δικαστήριο. Γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό χρειάστηκε μια δεκαετία. Κρεμεί στο δικαστήριο. Δεν έχει τελειώσει η υπόθεση αυτή. Μετά, τους μελλοντικούς πόρους γενικά και για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα ήθελα εγώ να έχουμε αρκετή χρηματοδότηση για τα κοινωνικά. Τώρα δεν ξέρω οτιδήποτε μπορεί να έχει ισχυριστεί, να μην έχει ισχυριστεί κάποιος πρέσβης. Και ο προπολογισμό είναι και η έκφραση ενός πολιτικού οράματος και μιας πολιτικής κατεύθυνσης. Και αν δείτε τον πυλώνα μας των κοινωνικών δικαιωμάτων με όλα αυτά τα μεγαλεπίβολα σχέδια και τις αρχέ μας, αυτά θα πρέπει να τα ελοποιήσουμε και αυτό χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Όχι μόνο νέα νομοθεσία ε, ε, που πρέπει εμεί να κάνουμε και να το κάνουμε, αλλά χρειάζονται και πολλές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Και καλούνται τα κράτη-μέλη να τις κάνουν. Εμείς μόνο υποστηρικτικά μπορούμε να τους βοηθήσουμε, αλλά ε, αυτό προϋποθέτει να έχουμε αρκετά χρήματα και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είμαστε ενώπιον μεγάλων αλλαγών, παγκοσμιοποίηση, ψηφιοποίηση. Θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα και ενέργεια να ενισχύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να είναι έτοιμοι για τη νέα οικονομία, για τους νέους τρόπους δουλειάς, να μην μένουν στην άκρη ή πίσω, αλλά και όταν είναι άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, να υπάρχει καλή υποστήριξη. Υποστήριξη δεν σημαίνει επίδομα. Δεν τι να το κάνω να παίρνει όλος επίδομα ανεργίας ή κάποιο άλλο προνοιακό επίδομα. Ε, δεν είναι αυτή η στήριξη. Χρειάζονται υπηρεσίες, χρειάζονται πραγματικές ε, δράσεις και αυτό εμείς θα ενθαρρύνουμε με τα δικά μας μέσα. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θέλουμε και καλό είναι να έχουμε και αρκετά χρήματα στον προπολογισμό για τα κοινωνικά για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιούμε ε, με ευελιξία όπου χρειάζονται περισσότερο για να δείξουμε και στους πολίτες ότι η Ευρώπη θέλει να τους βοηθήσει να αλλάξει η ζωή τους και να μην μείνει κανείς στην άκρη του δρόμου. Αυτό είναι ο, ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων, κυρία Πρόεδρε. Εσείς εγκρίνατε ένα χοντρό έγγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς βγάλαμε αυτό το φυλαδιάκι. Οι τρεις πρόεδροι των τριών θεσμικών οργάνων. Βάλτε το μαζί με το διαβατήριό σα και να το διαδώσετε παρακαλώ γιατί τα επόμενα χρόνια μας περιμένει πολλή δουλειά και στον προπολογισμό. Ευχαριστώ. Thank you very much. Sorry. Ευχαριστώ πολύ. Διαδικαστικό. Mm. Ναι. Ήθελα μόνο να πω, γιατί νομίζω ότι υπήρξε μια παρεξήγηση, ότι οι ερωτήσεις μου δεν ήταν εκτός ε, της ε, Επιτροπής. Ε, θέλουμε προπολογισμό απόδοσης, δηλαδή σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τους στόχους και την απόδοση του προπολογισμού. Είχα την εντύπωση πως νομίζατε πως οι ερωτήσεις μου δεν ήταν εντός του πλαισίου της Επιτροπής, ενώ ήταν. Όχι, όχι. Όχι, είναι αντίθετα το, το πρόβλημα ότι μπορούμε να μιλάμε για ώρες για τα θέματα της απασχόλησης ε, ενώ εδώ θα, και γι' αυτό είπα εδώ να μείνουμε μόνο στα θέματα του ελέγχου προπολογισμού γιατί αλλιώ θα κρατούσε για πάντα αυτή η συζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ γιατί φοβόμουν στην αρχή ότι δεν θα πάει καλά το πράγμα, γιατί Δευτέρα το απόγευμα είναι δύσκολη, δύσκολο, ε, γιατί όλοι φτάνουν τη Δευτέρα. Αντίθετα πήγε πάρα πολύ καλά η συζήτηση, φτάσαμε και σε φιλοσοφικά ζητήματα. Ευχαριστώ και δίνω και πάλι την Προεδρία στην Πρόεδρο Γκρέσλε. Συνεχίζουμε τη μέρησια διάταξη. Σημείο 4. Ein Bericht über unsere Missionsreise in Polen. Αποστολή της Επιτροπής ε, Κοντ στην Πολωνία. Τον Απρίλιο φέτος μετέβημεν στην Πολωνία. Δυστυχώς μόνο τέσσερα μέλη της Επιτροπής μας. Ο παρακαθήμενος συνάδελφος Βον, ο συνάδελφος Τσέλερ, ο συνάδελφος Τσερνέτσκι πήγαινε ερχότανε και μια άλλη συνάδελφος από την Πολωνία εκτός ποσοστώσεως και υποφαινομένη. Ενδιαφέρον το ταξίδι πρέπει να σας πω, όσο και σημαντικό. Είδαμε έργα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθωτικά ταμεία την έκθεση την έχετε ε, στους φακέλους σας. Ήταν πολύ μεγάλο το ταξίδι αυτό. Να εξετάσουμε λίγο την έκθεση. Αρχίσαμε στο Βρότσλαβ, ε, στο αεροδρόμιο που φτάσαμε όλοι, προσγειωθήκαμε εκεί. Έχει ανακαινιστεί με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τα βρείτε τα ποσά. Μετά πήγαμε σε ένα κέντρο τεχνολογίας και μετά είδαμε ένα υδραυλικό σύστημα. Στο Βρόσλαβ που είναι στο ποτάμι και συχνά πλημμυρίζει. Με πολλά εκατομμύρια βοηθήσαμε σε ένα σύστημα συγκράτησης των πλημμυρών εκεί φραγμάτων. Την άλλη μέρα πήγαμε στον αυτοκινητόδρομο που είδαμε μετά τα αντιπλημμυρικά και μετά πήγαμε στην Αρχιεπισκοπή ε, της Βαρσοβίας ε, σε ένα έργο της Αρχιεπισκοπής εκεί, ποιμαντικό και μετά είδαμε ένα αυτοκινητόδρομο. Ένα ΕΦΕ, e σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα λέω λίγο συγκεχημένα. Ναι. Εκεί στον αυτοκινητόδρομο. Μετά πήγαμε στην εταιρεία ε, Βίλτον. Έχουμε χρηματοδοτήσει εκεί ένα εργαστήριο για την αφαίρεση του θείου από ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ε, που χρηματοδοτήσαμε και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Το απόγευμα συζητήσαμε και πάλι τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Αν δείτε στο φάκελό σας, και θέλω να ευχαριστήσω τη γραμματεία που έχει κάνει τεράστια δουλειά από τη διοργάνωση μέχρι τη σύνθεση του φακέλου ολόκληρου. Αν δείτε λοιπόν στη σελίδα 22 ε, της έκθεσης ε, αυτό το πίνακα θα διαπιστώσετε τι έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μάλιστα έχει 85% χρηματοδότηση της κίνησης και βλέπετε πώς έχει η κυκλοφορία στην Πολωνία σε σύγκριση με τη Γερμανία και τη Γαλλία. Αυτή δεν ήταν δική μου ιδέα αλλά ήταν πολύ χρήσιμο από τη γραμματεία. Κοιτάξτε και την κίνηση. Έχουμε μεγάλες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Πολωνία, για σχετικά χαμηλή κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους, όχι παντού, αλλά 16.000, 17.000 τη μέρα οχήματα. Τίθεται ένα ερώτημα και ως συμπέρασμα. η επιλογή των έργων είναι πάντα τόσο εύστοχη. Και δεύτερον, είναι ευφυές να κινητοποιούνται δημόσιες επενδύσεις είτε πρόκειται για πλημμυρικά έργα, είτε πρόκειται για αυτοκινητοδρόμους και στην εταιρεία Βίλτον οι χρήστες και οι δικαιούχοι αυτή η εταιρεία που, είναι, που έχει φορτηγά έχει τώρα μεγάλα ε, γεμάτα ταμεία και έχει ε, εφορμήσει προς και, και, και κάνει αγορές και πολλές. Λοιπόν, ε, καλό είναι να χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια δημόσια έργα και να μην συμμετέχουν καθόλου οι χρήστες, οι τελικοί χρήστες ή δικαιούχοι. Γιατί όταν κάτι είναι δωρεάν δεν έχει και αξία τελικά. Ε, οι πολωνικές αρχές κάνουν καλή δουλειά, πραγματικά το είδαμε, το είπαμε και θα ήθελα να το επαναλάβω κι εγώ. Επίσης είδαμε ότι η Πολωνία ε, χειρίζεται μεγάλα ποσά, γιατί στα διαρθρωτικά ταμεία σε αυτή την περίοδο είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης. <laughs> Διαδέχθηκε την Ισπανία. Και είναι και μεγάλο το φάσμα των επενδύσεων που αποφέρουν καρπούς. Και η Πολωνία πραγματικά είναι στο δρόμο ώστε να γίνει μια σύγχρονη βιομηχανική χώρα. Έχει και εργατικό δυναμικό εκεί παρόν ε, και έχουν και ιδέες πώς να αξιοποιήσουν αυτά τα χρήματα. Οι περιφέρειες δεν είναι στραγγαλισμένες. Ε, ε, είδαμε το αποτύπωμα των επενδύσεων. Έχει αφήσει σημάδια η επένδυση και οι υποδομές που χρηματοδοτούνται και πραγματικά εξυγχρονίζεται, η Πολωνία έχει πιο σύγχρονη οικονομική διάθρωση και μου επιτρέψετε ένα πολιτικό σχόλιο. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο μεγάλη ατμόσφαιρα και κλίμα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέτοια απόρριψη ε, και επιφύλαξη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί τα λεφτά δεν πέφτουν από τον ουρανό είναι από φορολογουμένους άλλων κρατών, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία. Έρχονται λοιπόν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι, βάζουν το χέρι στην τσέπη, επενδύουν μαζικά στην Πολωνία και οι Πολωνοί θα επιθυμούσα αυτή η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εξυγχρονισμό της Πολωνίας να γίνεται αντιληπτή και κατανοητή και από τον πληθυσμό εκεί. Συναντήσαμε και το Εθνικό Ελεκτικό Συνέδριο και τη Βουλή, όπως πάντα, της Πολωνίας και είπαμε και εκεί ότι παρακαλούμε η Πολωνία να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και είναι σημαντικό για την προστασία ε, των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην μπαίνουν διαφορετικά κονδύλια και χρήματα χώρες που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε στην Πολωνία από την ένταξή της και καλό ήταν αυτό και σημαντικό και καλό θα ήταν να ξαναπάμε έτσι, σε κάποιο ορατό χρονικό ορίζοντα, γιατί είναι σημαντικό να ανακοινούμε κάποια ζητήματα ξανά και ξανά και να τα συζητούμε έτσι σε ένα επίπεδο και να τα προχωρούμε. Ε, πολύ ενδιαφέρον το ταξίδι, πάρα πολύ για μένα. Περίπου οργώσαμε τη μισή χώρα από το ένα έργο στο άλλο και οι συνάδελφοι που ήταν παρόντε και ο συνάδελφο Τσέλερ και ο συνάδελφο Βόν έχουν αποκομίσει εμπειρίε να μα πούνε δύο-τρία λόγια ε, για τι δικέ του απόψει. Ο κύριο Βόν. Yeah, yeah, Καλή σύνοψη αυτή, σαν να έχει περάσει πολύ καιρός, πολύ καιρός, ε, τον Απρίλιο νομίζω. Ε, αυτό που θυμάμαι είναι ότι ξυπνούσαμε νωρίς, και κοιμόμασταν αργά. Επίσης θυμάμαι ότι επισκεφθήκαμε πολλά έργα υποδομών, ό,τι υποδομές μπορείτε να το φανταστείτε. Οδικές μεταφορές, αεροδρόμιο, σιδηροδρόμους, ε, ε επεξερασίας ύδατος. Πάντα επισκεπτόμαστε ε, εργοστάσια επεξερασίας υδάτων τα περισσότερα από αυτά τα έργα ήταν καλά, δεν νομίζω ότι εντοπίσαμε κάποια απάτη. Δεν με ανησυχεί το θέμα αυτό. Το μόνο που μας ανησύχησε λίγο ήταν στον καθεδρικό του Ρόσλαβ. Αρκετά εκατομμύρια λίρες αφιερώθηκαν σε αυτό το project το οποίο δεν αύξησε πολύ την επισκεψιμότητα του καθεδρικού. Ε, δεν είμαι σίγουρος για την αποδοτικότητα αυτής της χρηματοδότησης. Δεν λέω να μην χρηματοδοτούμε τέτοιου πολιτιστικά έργα στο μέλλον, αλλά θα χρειαστεί να έχουμε περισσότερη καλύτερη αιτιολόγηση. Ε, νομίζω θα πρέπει να το δούμε αυτό ε, την επόμενη προγραμματική περίοδο μετά το 2020. Κύριε Στέλλερ, δυστυχώς δεν συμμετείχα, δεν μπόρεσα να συμμετάσχω αυτή την προσωπία, αλλά επειδή έχω γεννηθεί στη Σιλεσία, ε, αισθάνομαι πολύ κοντά στη γειτονική μας χώρα και παρακολουθώ πάρα πολύ προσεκτικά και στενά τις εξελίξεις και συχνά πηγαίνω στα μέρη που επισκέφθηκε η αντιπροσωπεία. Θα ήθελα λίγο να προειδοποιήσω για το σημερινό κλίμα που καλλιεργεί η σημερινή κυβέρνηση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην νομίζετε ότι αυτό ισχύει για όλη τη χώρα, ούτε για όλο το λαό. Αν πάτε στο Βρόσλαο, πήγατε στο, στο Βρόσλαο, ε, Μπρέσλαου στα γερμανικά, θα δείτε ότι ο Δήμαρχος είναι πάρα πολύ ευρωπαϊστής, είναι υπέρ της ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης, πάγια στο παρελθόν. Πέρσι μάλιστα ήταν το Βρόσλαφ πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και είναι απέναντι στη γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση της Βαρσοβίας. Ακόμα και το 2008 όταν όλα τα κράτη μαζί με τη Γερμανία είχαν αρνητική ε, οικονομική ανάπτυξη, η Πολωνία είχε θετική. Πράγμα που επηρέασε και τα διορθωτικά ταμεία και την επιρροή τους. Και σε αυτά οφείλεται άλλωστε ότι ε, κατάφεραν να δημιουργήσουν και ανάπτυξη και απασχόληση το θέμα για τις υποδομές και συγκοινωνιών. Σημερίζομαι την κριτική της Προέδρου. Βεβαίως ε, χτίστηκαν αυτοκινητόδρομοι. Γιατί ε, ε είχαν ε, ε, το παγκόσμιο πρωτάθλημα να διοργανώσουν το Μουντιάλ, αλλά είναι το τοπίο έτσι, πάρα πολύ, καμιά φορά μονότονο και ανιαρό ε, για τον οδηγό. Επίσης με ευρωπαϊκά κονδύλια αγοράσανε κάτι περιπολικά υπερσύγχρονα για την αστυνομία με όργανα μέτρησης κτλ. Επίσης υπήρχαν και κάποια εκατομμύρια ειδείς που πήγαιναν στο σιδηρόδρομο και τελικά κατέληξαν στον αυτοκινητόδρομο. Έχουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα για τη σύνδεση των κρατών της Βαλτικής μέσω Πολωνίας με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά στο μεταξύ ε, έχει σταματήσει η σιδηροδρομική σύνδεση ε, Πολωνίας-Λιθουανίας γιατί δεν επιτρέπεται πια να κυκλοφορεί ένα τρένο με ταχύτητες 30 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή είναι το δίκτυο τέτοιο που δεν αντέχει. Ε, άρα θα πρέπει τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιούνται και για ένα ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Κατά τα άλλα, το είδαμε και το Σαββατοκύριακο, πολλοί άνθρωποι στο δρόμο της Πολωνίας. Η Πολωνία παραμένει ένα σημαντικό μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις των ανθρώπων και ξέρουν να εκτιμούν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η κυρία Πιτέρα, παρακαλώ. <clears throat> Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι βουλευτής από την επαρχία Μαζοβιέσκη, ε, ακόμα και αν στην Βαρσοβία. Αυτή είναι η εκλογική μου περιφέρεια. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την ε, περιοχή και επισκέπτομαι πόλεις και χωριά τακτικά. Γνωρίζω πόσο καλά χρησιμοποιούνται οι, ε, τα ταμεία. Η περιφέρεια αυτή έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και εγώ παρακολουθώ εκ του σύνοικης τις εξελίξεις ε, ως Ευρωβουλευτής. Ε, όντως υπήρξαν προβλήματα σε επίπεδο υποδομών. Μιλώ για τον αυτοκινητόδρομο και μπορώ να σας πω ότι αυτοκινητόδρομο στην περιφέρειά μου <coughs> είναι εξαιρετικά φορτωμένοι. Ίσως αυτό το κομμάτι του δρόμου S8 σε 5 με 10 χρόνια να χρησιμοποιείται ε, και ακόμη περισσότερο διότι ε, γίνονται μεγάλες ε, δημογραφικές μετακινήσεις στην Πολωνία όσον αφορά την κατοικία των ανθρώπων, οι οποίοι μετακινούνται πολύ και πιστεύω πως έτσι θα εξισυρωπηθεί η χρήση του αυτοκινητοδρόμου αυτού και των δρόμων γενικότερα. Τώρα όσον αφορά τον ευρωσκεπτικισμό, στην πραγματικότητα οι Πολωνοί είναι υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πρόβλημα για μένα ως Ευρωβουλευτή αλλά και για τους υποστηριχτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αυτός ο ευρωσκεπτικισμός εκφράζεται από την ίδια την κυβέρνηση ενώ τα στοιχεία μας δείχνουν το 80% των ε, Πολωνών πολιτών είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι θετική. Και περνάμε δύσκολους καιρούς, όμως οι Πολωνοί πολίτες ε, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από τα χρήματα εγγυάται την ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ναι, το καταλαβαίνουμε και μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση αυτή. Κανείς δεν επιθυμεί μια τέτοια κατάσταση και αποδυναμώνει και τη χώρα. Μια χώρα που είναι τόσο διχασμένη θα έχει συνέπειες και για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από τη Γενική ε, Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θέλω να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μην διστάσετε να μας πείτε τι ξεχάσαμε και πρέπει να ξανακοιτάξουμε. Euh, madame la Présidente. Δύο λόγια για την έκθεση, πολύ καλή κατά τα άλλα. Συμφωνούμε με τα συμπεράσματα σε μεγάλο βαθμό. Να σχολιάσω κάποια από αυτά που είπατε στην εισαγωγή σας. Πρώτον, για την μειωμένη κίνηση σε, ορισμένες, σε ορισμένους Στη σελίδα 22 έχει, υπάρχει ένας πίνακας με συγκεκριμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων και που συγκρίνει με αντίστοιχες υποδομές στη Γαλλία και τη Γερμανία. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε εμείς στην Κομισιόν για την αξιολόγηση ενός σχεδίου όταν αυτό είναι πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας, ε, η μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι ε, η ανάλυση της ε, ε, οικονομικής αποδοτικότητας που, σχετίζει, που συσχετίζει την επένδυση με την χρήση του, της υποδομής. Οπότε αυτά τα έργα είναι ένα κομμάτι αυτών στα οποία αναφέρεστε εσείς και σε κάθε περίπτωση η ανάλυση αυτών των συγκεκριμένων υποδομών είχε δώσει θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή η επένδυση ήταν αιτιολογημένη. Σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια, εκ των υστέρων ε, παρατηρήθηκε ότι η ε, πραγματική κίνηση ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη και αυτό ελήφθη υπόψη στην αξιολόγηση των επόμενων σχεδίων. Δεύτερον, ε, η συμμετοχή των χρηστών σε ορισμένες επενδύσεις κάτι που σχετίζεται και με ένα συμπέρασμά μας, συμπέρασμά σας για την ε, βιωσιμότητα ε, των υποδομών αυτών, δηλαδή το γεγονός του κατά πόσον, την ερώτηση του κατά οι χρήστες μπορούν να αγγιθούν την ε, λειτουργία αυτών των υποδομών στο μέλλον. Η, τα μια ταμεία κατανέμουν τις αρμοδιότητες κατανέμουν την χρηματοδότηση ε, μεταξύ ε, της κρατικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης αφενός και την συμμετοχής των χρηστών αφετέρου. Όμως, η Κομισιόν δεν επιβάλλει στα κράτη-μέλη κάποια τιμολογιακή πολιτική. Ορισμένα κράτη πράγματι ε, μειώνουν πάρα πολύ τις χρεώσεις προς τους χρήστες και τους μολύνοντες. Ε, την περίοδο 2014-2020 είχε αποφασιστεί να εφαρμόσει τη αρχή του ορυπαίνων πληρώνει και με αυτόν τον τρόπο χρεωνόντουσαν μεγαλύτερα ποσά στους χρήστες. χρήστες. Η συμμετοχή των χρηστών αυξήθηκε διότι ζητούμε οι χρήστες να καλύπτουν ε, και την απόσβεση και τρίτον ε, όταν οι χρήστες δεν είναι ερυπαίνοντες, για παράδειγμα χρήστες υποδομών δημόσιων μεταφορών ε, ή πολιτιστικών υποδομών τότε για παράδειγμα το Μπρότσλαου ήταν αυτό, τέτοια περίπτωση τότε. Η ελαστικότητα της ε, ζήτησης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με τρόπο πιο λεπτό προκειμένου η αύξηση των εισιτηρίων, των διοδίων κλπ. να μην οδηγεί στη μειωμένη χρήση της υποδομής. Υπάρχουν αδυναμίες αλλά οι κανόνες του 2014, της περίοδου 2014-2020 έχουν ενισχυθεί πλέον για να αυξηθεί η συνεισφορά των χρηστών. Δεν ξέρω αν η συνάδελφός μου από τον έλεγχο, δημοσιονομικό έλεγχο θέλει να πει κάτι. Ε, good afternoon, ladies. Είμαι η ε, επικεφαλής της ε, μονάδα ελέγχου τη Γενική Διεύθυνσης Ρίτζιο. Θέλω να πω το εξή. Σε ό,τι αφορά την απλοποίηση και την ε, υπερ, νομοθετική υπερφόρτωση, να σας πω το εξή. Στην περίοδο 2014-2020 εξετάσαμε τέτοιου είδου περιπτώσεις των ε, ε, υπερθεματισμών, υπερθεματισμό, νομοθετικό υπερθεματισμό. Βρήκαμε κάποιες περιπτώσεις, οι οποίε έχουμε ε, αναφέρει. Έξι υποστολές έγιναν στην ε, Πολωνία που αφορούσαν τη διαχείριση και την επιλογή των σχεδίων και σε ό,τι αφορά το πόρισμά σας για τις περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες επιλογής, το επιβεβαιώνουμε. Θα το δείτε όταν δημοσιευθεί η έκθεσή μας. Αυτό παίρνει 9 με 12 μήνες καμιά φορά. Συγγνώμη, η διαδικασία επιλογή σχεδίων παίρνει 9 με 12 μήνε πολλέ φορέ. Δεύτερον, για την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ, κατά τη διάρκεια των εργασιών ε, εκαθάρισης ε, θα μεριμνήσουμε έτσι ώστε ο ΦΠΑ πραγματικά να αφαιρεθεί. Μάλιστα. Μια ερώτηση να σας κάνω. Από τους αριθμούς που έχουμε μας δημιουργήθηκε και η εντύπωση ότι από πλευρά διαχείριση θα πάνε πολύ καλά οι Πολωνοί. Τη συμμερίζεστε αυτή την άποψη. Ε, Όσον αφορά την ε, ε, γεωγραφική περιφέρεια και τις επαφές που έχουμε καθημερινά σχεδόν με τις πολωνικές αρχές επιβεβαιώνω αυτό που είπατε ότι η συνεργασία είναι καλή εμείς ε, ε, σε εκθέσεις της Όλαφ και από τους ελέγχους που ε, διεκπαιρεώσαμε ήδη δεν έχουμε φόβους όσον αφορά τις δαπάνες και εν γέννη συνεργασία γίνεται σε επικοδομητικό πνεύμα, δηλαδή προτάσεις της Κομισιόν περί της διαχείρισης και ειδικά για το θέμα της απλοποίησης που είναι μία από τις βασικές μας ανησυχίες αυτή τη στιγμή ε, μας επιτρέπει να έχουμε κανοποιητικά αποτελέσματα. Επιβεβαιώνουμε λοιπόν την ποιότητα της σχέσης ε, με τις αρχές. Ε, just Επιπλέον, να συμπληρώσω από την άποψη του ελέγχου ότι συνεργαζόμαστε στενά με την ελεκτική αρχή και έχουμε τακτικές ε, συνεδριάσεις για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα της ελεγκτικής μας εργασίας. Αυτή τη στιγμή κάνουμε επιλεκτικές επιχειρήσεις και έλεγχο της διοίκησης. Η Όλαφ έχει κάνει λοιπόν αυτή τη συνεργασία ώστε να ελέγχουμε ε, σε ένα πρώιμο στάδιο και αν υπάρχουν ζητήματα να προχωρήσουμε και σε πιο εις βάθος ελέγχους. Αλλά η εργασία του ελέγχου είναι ήδη αξιόπιστη και πάνε, πάνε τα πράγματα καλά λοιπόν ομαλά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε αυτό το σημείο στη Μέση Διάταξη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και για όλους τους παρόντες ε, στην ε, αντιπροσωπεία. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εκεί. Για τόσο μεγάλα κράτη Καμιά φορά ε, θα ήθελα να είναι πολυπληθής η αντιπροσωπεία. Τουλάχιστον ε, όσο με την Ουάσιγκτον και έχουμε περάσει στο επόμενο θέμα. Για πρώτη χώρα, μετά από καιρό, επτά συνάδελφοι μετέβημεν εκεί. Η συνάδελφο Σμιτ που είναι παρούσα, είχε έρθει μαζί και παρακαλώ να συμπληρώσετε τα όσα θα, θα πω. Ποιο ήταν ο στόχος του ταξιδιού αυτού που είχε αναβληθεί πολλά χρόνια με πολλές αμφιταλαντεύσεις, τελικά έλαβε χώρα. Να δούμε το αμερικανικό σύστημα που έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί έχουν πολύ υψηλό ποσοστό σφάλματος, 10%. Και θέλω να δούμε τι μετράνε και πώς τα κάνουν εκεί αυτά τους ελέγχους. Πριν από λίγα χρόνια, το παλιό κοινοβούλιο είχε κάνει συνεδρίαση της Επιτροπής μας και εργαστήριο. Είχαμε προσκαλέσει ε, Αμερικανούς και είδαμε ότι τα στήματά μας διαφέρουν πάρα πολύ. Αυτή τη φορά ασχοληθήκαμε και με την κατάρτιση του προπολογισμού αλλά και πόσο στοχευμένος είναι ο προϋπολογισμός και πόσο συγκεκριμένος και ακριβής και ποιες είναι οι δυνατότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου, πώς δουλεύει το ελεγκτικό συνέδριο και κυρίως αξιοποίησαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με διεθνείς εταίρους της Ένωσης, όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Πήγαμε και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να δούμε τη συνέχεια που δίνουν στο θέμα της IT ε, τι διαπιστώσαμε λοιπόν, ότι οι Αμερικανοί με όσες διαφορές και αν έχει το σύστημά τους έχουν συνηθίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τους τραβάνε και τα αυτιά. Συμμετείχαμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονομικών, της Ομόλογης Επιτροπής, και εκεί τους ανέκριναν κανονικά. Δεν θα ήθελα καθόλου να είμαι στη θέση τους, αυτός που, που ήρθαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις της Επιτροπής. Ε, με πάρα πολύ στοχευμένες ερωτήσεις, συμπληρωματικέ ερωτήσεις, εκεί χωράμε η βελτίωση η δικιά μας Επιτροπή. Μετά, ε, τι άλλο είδαμε, ότι οι Αμερικανοί ε, ποντάρουν πάρα πολύ στον εσωτερικό έλεγχο και με γενικούς επιθεωρητές που έχουν και πολύ προσωπικό. Η Γενική Επιθεώρηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης μας υποδέχτηκε που έχουν χιλιάδες υπαλλήλους γιατί ελέγχουν δικαστήρια, σοφρονιστικά καταστήματα, δικαστήρια και η Γενική Επιθεώρηση έχει και αστυνομικές ε, ε, όπως το FBI. Μπορεί να κάνει και έρευνες αλλά και συλλήψεις το ίδιο. Έχει αρμοδιότητες δηλαδή ε, FBI, περίπου όλα ε, ο Γενικός Επιθεωρητής, ο εσωτερικός, ε, οικονομικός. Ε, και αυτά τα συστήματα μας έδειξαν πόσο εξαρτώνται από την πολιτική σε μια κρίσιμη φάση πολιτικά για την ε, Αμερική. Αν θεωρεί καλό ο πρόεδρος να τους απολύσει όλους, τους απολύει. Δεν έχει κανένα θέμα. Συλλήβδη. Äh, Καταλαβαίνετε ο πρόεδρος τι εξουσία έχει και στα ελεκτικά συστήματα και πώς μπορεί να τα καταργήσει και πώς μπορεί και να τα στήσει έτσι ώστε να μην γίνεται κανένας έλεγχος. Αυτό ήταν προφανές για όλους τους ε, συμμετέχοντες και έχουμε εκεί μια διαλκυστίδα μεταξύ του Προέδρου και διαφόρων κρατικών αρχών ενδιαφέρουσα και το συζητήσαμε ε, με ανθρώπους που είναι σήμερα σε θέσεις κλειδιά και το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, τουλάχιστον εγώ. Πήγαμε και στο Λευκό Οίκο, στον αρμόδιο εκεί διευθυντή για τον προπολογισμό, που εκείνη τη μέρα είχε καταθέσει τον προπολογισμό του στη Γερουσία και στο μεταξύ ε, του το κάνανε πραγματικά ε, φίλο και φτερό. Με καθόλου επαγγελματικό τρόπο πρέπει να πω καταρτίζεται. Ναι, καλά, πώς να το πω τώρα το, με, ποιο τρόπο φτιάχνουν τον προπολογισμό δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι καταρτίζεται με το σωστό τρόπο. Ήταν ενδιαφέρον το ταξίδι. Ένα, ε, μια μέρα αφιερώσαμε στην Παγκόσμια Τράπεζα, είχαμε διαφόρους αρμοδίους εκεί και μας εξήγησαν και το εσωτερικό ελεγκτικό σύστημα επιθεώρηση της ε, Παγκόσμιας Τράπεζας και σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον επαναλαμβάνω ε, το ότι προσπαθεί σε διάφορα επίπεδα η Παγκόσμια Τράπεζα να εφαρμόσει το θέμα της δεοντολογίας και της ηθικής και με πολύ μεγάλες υποχρεώσεις για τους υπαλλήλους και για εκείνους που δρούν εξ ονόματος για τα οικονομικά συμφέροντα. Και με ποια συνέπεια λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και εμείς υπολοιπόμεθα. Για την IT, γιατί μας απασχόλησε αυτό το θέμα, ε, συζητήσαμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βέβαια, ένα τμήμα της επίσκεψης είχε να κάνει και με πολλές αναμονές ε, για θέματα ασφαλείας, ελέγχους ασφαλείας και διεκπαιρέωσης. Καλό είναι να το συζητήσουμε αυτό το θέμα της IT κάποια φορά, γιατί δεν έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση, πόσο μάλλον θετικά από το σεισμό του 2011 και την τότε επίσκεψή μας για τα μέσα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτά είχα να πω εγώ. Ενδιαφέρουσα η επίσκεψη αυτή για να δούμε πώς λειτουργούν οι διάφορες υπηρεσίες και τι δυνατότητες έχουν και η πραγματική αξία και η υπεραξία ήταν ότι πρέπει να μεταξελίξουμε και τα δικά μας συστήματα και να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Για να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στη δράση μας κύριε Τσέλερ και κυρία Σμιτ που ήσασταν στην επιτροπή μας εκεί. Θέλετε να συμπληρώσετε τίποτα. Με Με Ευχαριστώ. Τι να συμπληρώσω. Τα είπατε όλα. Ε, το ενδιαφέρον ε, που μας έκανε μεγάλη εντύπωση εμείς κάνουμε μια δουλειά για να βελτιωνόμαστε πάντα και είδαμε και ένα προϋπολογισμό που δεν είχε ακόμα ε, εξαντληθεί και πώς γίνεται η συζήτηση. Όχι, ε, οι περικοπές δεν είναι με βάση τις, επιθυμι... με... βάση τις εμπειρίες ή τις ανάγκες, αλλά βγάζει φυρμάνια ο πρόεδρος. Αυτό θα περικοπεί, αυτό θα κοπεί τελείω, αυτό θα αυξηθεί και αυτό δεν χρειάζεται. Δεν έχει καμία σημασία τι είπε ο έλεγχος και τι διαπίστωσε. Αν θεωρεί ο πρόεδρος ότι πρέπει να γίνουν περικοπές, γίνονται. Και δεν πάει να είστε οποιοδήποτε οργανισμός αρχίζει γενομένης από τους βετεράνους, που βέβαια δεν τους κόβουν τα λεφτά, αλλά ο καθένα κανονίζει την πορεία του γιατί αποφάσισε ο πρόεδρο έτσι με, με φυρμάνει να κοπήμουν τα λεφτά. Αυτά και μέσα στο, στο μέλλον χρειάζονται άλλοι. Α, και ο ξενάδελφο Πυρίσκη ήταν παρόν, συγγνώμη. Το είχα ξεχάσει. Παρακαλώ. That's okay. Uh, thank you. Δεν, ε, ναι, ευχαριστώ. Πιστεύω πως ήταν ε, μια Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σειρά συναντήσεων που είχαμε στη Washington που μας ε, προβλημάτισαν και μας έδωσαν τροφή για σκέψη. Είχαμε full πρόγραμμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και με τις διάφορες επιτροπές και τη κυβέρνηση πολύ καλά διοργανωμένο πρόγραμμα. Ως προς την ουσία, και τη διαφορά περιθωρίου σφάλματος ανάμεσα σε εμά και το 10% που χρησιμοποιείται ως ε, κατόφλι στη ΣΥΠΑ. Να τονίσουμε και αυτό που αναφέρθηκε στα πορίσματα, πως το γενικό, Γενική Υπηρεσία Λογαριασμών δεν, ε, ε, δεν μετράει το ποσοστό σφάλματος ε, ε, φόλης της ύλης, αλλά κάνει, ένα, κάνει τους λογαριασμούς, ε, βγάζει ένα δελτίο ανά οργανισμό και αυτό είναι πιο ευέλικτο και μόνο όταν επί τρία συναπτά έτη ξεπερνιέται το περιθώριο σφάλματος εκδίδεται σχετική προειδοποίηση από το αρμόδιο γραφείο και έπειτα δεν υπάρχει διαδικασία απαλλαγής της ΣΥΠΑ και αυτό το οποίο τονίζουν ε, όμως ε, στις εποπτικές επιτροπές είναι ακροάσεις. Ακροάσεις, ε, στη μία ήμασταν και παρόντες και είχε να κάνει με τις πρακτικές τις ευημερίες όσον αφορά τη χρηματοδότηση των φοιτητών. Βεβαίως έχω Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση του κοινού σε αυτές τις δημόσιες ακροάσεις και το Ευρωκοινοβούλιο θα μπορούσε να σκεφτεί νομίζω τρόπους ώστε να αυξήσει, μάλλον να τονώσει αυτό το δημόσιο μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στο κοινό. Αυτό που προσπαθούμε εξάλλου να κάνουμε, να αυξήσουμε δηλαδή την ενημέρωση και να δείξουμε τις κακές πρακτικές. Κάτι ακόμα που πιστεύω ότι αξίζει να αναφέρουμε είναι το γεγονός ότι όπως είπαμε, το σύστημα των γενικών επιθεωρητών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το Υπουργείο Γενικών Υποθέσεων, όπου έχει έναν συγκεκριμένο διευθυντή και 15 χρόνια, έχει πολύ, χέρι μεγάλης προστασίας από το Κογκρέσο. Προστατεύεται δηλαδή από την πολιτική επιρροή και χειραφετείται σε εντυπωσιακό βαθμό για να κάνει τη δουλειά του ανεξάρτητα και αμερόληπτα. Κάτι ακόμα είναι ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται και τον ίδιο τον προπολογισμό, τον ομοσπονδιακό προπολογισμό, όπου μάθαμε ότι εστιάζουν την προσοχή σε ένα τέταρτο του προπολογισμού, το οποίο μπορούν να επηρεάσουν και που αφορά τρέχουσες αποφάσεις. Επίσης το Κογκρέσο ε, εκφράζεται επί του προϋπολογισμού και προβαίνει σε διαπραγματεύσεις με το εκτελεστικό, με την κυβέρνηση. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό είναι ότι όντως ενδιαφέρονται για το ποσοστό μεγέθυνσης, όχι τόσο για το έλλειμμα ή το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ και αυτή είναι διαφορετική προσέγγιση από αυτήν που έχουμε εμεί εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή τη μανία που έχουμε με τη λιτότητα. Θα πρέπει να πω ότι η αμερικανική προσέγγιση φαίνεται να αποδίδει καλύτερα. Και μια από τις πτυχές που προέκυψαν επίσης είναι ότι βασικά εστιάζονται στις επιδόσεις και όχι στη συμμόρφωση όταν ε, εξετάζουν τη λειτουργία του προπολογισμού. Τέλος, ο κ. Βέιν ε, μας είπε σαφώς ότι θα κάνουν ανταγωνισμό στη φορολογία με την Ευρώπη. Και αυτό θα πρέπει ίσως να το σημειώσουμε, αξίζει τον κόπο. Ευχαριστώ. Μάλιστα. ενδιαφέρον. Ο Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όσο το δολάριο είναι παγκόσμιο απόθεμα ως νόμισμα, δεν χρειάζεται ε, να σκέφτονται το χρέος, μπορούν να αυξήσουν τα επιτόκια και θα πληρώσει ο κόσμος το χρέος. Και μπορούν να έχουν 40 δις ε, το μήνα έλλειμμα εμπορικών συναλλαγών. Εγώ δεν μπόρεσα να συμμετέχω, είχαμε και άλλες αντιπροσωπείες γιατί είναι πάντα σε πράσινες εβδομάδες. Γι' αυτό με ενδιαφέρει πολύ αυτό που είπατε ότι ήσασταν και στην Παγκόσμια Τράπεζα πήγατε. Είναι είναι έδρα πολλών διεθνών οργανισμών που χρηματοδοτούνται γενναία από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Βλέπε Παγκόσμια Τράπεζα. Και συχνά όταν θέλουμε να μάθουμε αν τα λεφτά μας έπιασαν τόπο ε, και τα προγράμματα που χρηματοδοτούμε για την υλοποίηση στην αναπτυξιακή βοήθεια μέσω της τράπεζας είναι πάρα πολύ φιδωλή στην πληροφόρηση. Δημερώς δεν μπορούμε να το δούμε αυτό με την Παγκόσμια Τράπεζα να μας ενημερώνουν για το πώς χρησιμοποιούν τα κονδύλια που τους δίνουμε εμείς στα προγράμματά τους και τι επίπτωση έχουν και τι αντίκτυπο. Μετά ο ΙΕ με τις διάφορες υπηρεσίες του και αυτός χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο που η ίδια δεν είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών παρά μόνο τα κράτη-μέλη της. Είμαστε ο βασικός ε, χρηματοδότης πολλών οργανισμών του ΟΗΕ. Μήπως να ζητήσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στην εκταμείευση των πόρων. Να πιέσουμε κιόλα ε, για τις οργανώσεις του ΙΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση έγινε τίποτα. Είχατε καμία συνομιλία. Που να έχει και αποτελέσματα για μας. Yeah, Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά. Γι' αυτό το λόγο πήγαμε άλλωστε εκεί. Και οπωσδήποτε στην υποχρέωση λογοδοσίας μπορούμε να κάνουμε κάτι όλη η Επιτροπή μας. Ναι. Α, για την ΑΕΤ ξέχασα να πω ο κ. Τσέλερ, το Δεκέμβριο η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται θα συνεδριάσει στην ΑΕΤ. Αν υπάρχει καμιά ενημέρωση που μπορούμε εκεί να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε, θα σας ήμουν ευγνώμων. Με χαρά. Η έκθεσή μας... Αυτό, τι μάθαμε από το Δούνου του, ότι τα διαρθωτικά προβλήματα παραμένουν στο ακέραιο. Από το 2011 δεν έχουν αλλάξει πολλά, όσο μάλλον έχουν βελτιωθεί. Η κυρία Πύρης από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού. Thank you, um, Ευχαριστώ. Ελπίζουμε ότι ήταν ευκαιρία να μάθουμε από την Παγκόσμια Τράπεζα και να συνεργαστούμε στο πλαίσιο της ε, συμφωνίας πλαίσιο που έχουμε με την Παγκόσμια Τράπεζα. Είχατε την ευκαιρία να δείτε την ε, πλατφόρμα δωρητών που είναι ένα πραγματικό πολύ καλό εργαλείο διαφάνειας ε, σε πραγματικό χρόνο. Ε, είναι κάτι το οποίο, στο οποίο έχουμε συνεργαστεί με την Παγκόσμια Τράπεζα. Ναι, ακριβώς, πράγματι. Είχαμε ενδιαφέρουσες συναντήσεις εκεί όλη μέρα. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η Παγκόσμια Τράπεζα είναι υπόλογη σε εμά, αλλά είναι και πολύ ειλικρινής και με χαρά το κάνουν και αν υπάρχουν ειδικά έργα που έχετε υπόψη σας να μας τα πείτε για να ε, προετοιμάσουμε την ερώτηση αυτή. Λοιπόν, ολοκληρώνεται και αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη, καθώς και η δημόσια συνεδρίασή μας και παρακαλώ να αποχωρήσουν όλοι όσοι δεν έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στην κεκλεισμένη των θυρών συνεδρίαση. Ή δυνατόν αθόρυβα όσο και γρήγορα. Und dann möchte ich auch das Konsekretariat bitten zu checken. Και παρακαλώ τη γραμματεία να τσεκάρει αν πραγματικά αποχωρούν όσοι δεν έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται.